Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι γιατί η ατζέντα μας είναι υπερπλήρης και έχουμε και καλεσμένους. Mm. Γι' αυτό θα αρχίσουμε με το σημείο 8 της σημερινής διάταξης του Κοινό Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων και η συγκέντριά μα είναι η κυρία Μαριάν Τάισεν και τη δίνω μέσα στο λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω του που κατέθεσαν ε, τροπολογίες. Αυτά είναι υλικά που μοιάζουν απλά για τους οικονομολόγους, αλλά είναι δύσκολα για τους δικηγόρους. Οπότε χαίρομαι για το ότι τόσο πολλοί κόσμος έκανε προσπάθειες ε, να βελτιώσει αυτή τη γνωμοδότηση που πρέπει να πάει στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Γιατί όλα αυτά νομίζω μπορούν να μας βοηθήσουν και να δώσουμε έτσι μια καλύτερη γνωμοδότηση. Βεβαίω υπάρχει μια εξαίρεση, είναι μια τροπολογία του ECR. Η πρόταση αυτή αφορά το διασυνοριακό εμπόριο το οποίο πρέπει να προωθηθεί για να βοηθηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και να γίνει με έναν τρόπο που θα είναι νομικά απλός. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια Όποιος έχει τώρα κάτι ενάντια σε αυτή την, την πρόταση, εντάξει, μπορεί να πει πως μπορεί να, να βελτιωθεί. Και προς ε, αυτή την κατεύθυνση νομίζω συμβολεύουμε την νομική επιτροπή. Οπότε για τη συγκεκριμένη αυτή τροπολογία εγώ θα είμαι αρνητική. Κατόπιν υπάρχουν τρεις τροπολογίες ε, που αφορούν ε, αφενός ε, την προσαρμογή σε σχέσεις B2B μεταξύ επιχειρήσεων. Πάνε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν τροπολογίες λοιπόν που θέλουν να βγάλουν αυτό το κομμάτι από την πρόταση της Κομισιόν και άλλες λένε πως τα B2B πρέπει να αφορούν και μεγάλη επιχείρηση με μικρομεσαία επιχείρηση και δύο μεγάλες επιχειρήσεις. Τα διάβασα εγώ πάρα πολύ καλά και τις τροπολογίες και μπορώ να προτείνω να μείνει εκτός το B2B, να μην το στηρίξουμε γιατί θεωρώ ακριβώς πως ε, θα δώσουμε ειδική μεταχείριση στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει βέβαια και η αρχή Think Small First και νομίζω πως ταιριάζει αυτό με την προσέγγιση μας. Οπότε πρέπει να το αφήσουμε μέσα γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν την ίδια δύναμη με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μετά υπάρχει η πρόταση Βενγκίγκολτ να ισχύσει αυτό για όλες τις επιχειρηματικές συμβάσεις και μπορώ να συμφωνήσω γιατί επειδή λέμε Think Small First δεν σημαίνει αποκλειστικά για τις μικρόμεσες επιχειρήσεις, γιατί αν και οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτή την Ευρωπαϊκή Σύμβαση και με τις μεγάλες επιχειρήσεις και με τις μικρομεσαίες, τότε καλό θα είναι, μπορούν να προσαρμόσουν περισσότερα, περισσότερα τα πράγματα, θα υπάρξουν ευκολότερα και γρηγορότερα ερμηνείες και θα ενηλικιωθεί το σύστημα αν θέλετε γρηγορότερα. Οπότε μπορώ να στηρίξω την πρόταση Sven Giegold. Τρίτη σειρά τροπολογιών που αφορά την ρήτρα αναθεώρησης ή αξιολόγησης αν θέλετε. Με κάποιες από αυτές μπορώ να συμφωνήσω και εγώ έχω καταθέσει τροπολογίες για τα ζητήματα που πρέπει να εξετάζουμε όταν θα γίνει, παράδειγμα, χάρη μετά από δύο χρόνια πρώτη αξιολόγηση και κοιτάζοντας τις τροπολογίες των συναδέλφων δεν έχω πρόβλημα με την τροπολογία 19 και 18 που ζητάνε να υπάρξει ένας βαθμός ε, αποδοχής ε, ο οποίος θα πρέπει να ερευνηθεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και από όλες τις επιχειρήσεις Οπότε συμφωνώ. Επίσης, να εξάζουμε το εάν θα οδηγηθούμε σε χαμηλότερο κόστος συναλλαγών και εδώ πέρα συμφωνώ με τον κύριο Πρεσέντε. Μετά υπάρχει η τροπολογία 11 του κύριου Γκίγκολτ που ζητάει να πάμε και σε πιο πολύπλοκα προϊόντα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειας. Θα προτιμήσω να μην πάω σε αυτό το θέμα. Είναι τόσο ειδικέ αυτές οι υπηρεσίες που έχουν δική τους νομοθεσία και αντιλαμβάνομαι πως και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή προετοιμάζει ένα προαιρετικό μέσο που θα αφορά τα ασφαλιστικά συμβόλαια. Επίσης υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο ε, χρεοκοπίας ε, και άλλες προτάσεις οι οποίες πάνε πάρα πολύ μακριά αλλά βεβαίως είναι αναγκαίο η ρήτρα αναθεώρησης ή αξιολόγησης να επεκταθεί και με κανόνες που ε, αφορούν την αδικοπραξία. Το έχω βάλει και σε ένα εκτιμώντας και συμφωνώ και με την πρόταση του κύριου Γκίγκολτ. Μετά έχουμε τροπολογία 20 του συναδέλφου Πρεσέντο που συνδέεται και με άλλες. Μπορούμε να βρούμε νομίζω ένα συμβασμό εδώ πέρα. Μετά υπάρχει ε, άλλο ένα πακέτο που αφορά τις ασφάλειες που είναι συνδεδεμένες με την αγορά αγαθών. Συμφωνώ με αυτή την ανησυχία και συμφωνώ πως η ιδιαιτερότητα των ασφαλιστικών συμφωλέων σημαίνει πως εδώ πέρα πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό νομοθετικό καθεστώς, αλλά αποκλείεται του χάρη όταν μιλάμε για σχετικές υπηρεσίες να μην αναφέρονται και οι χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε, οπότε συμπεριλαμβάνονται εδώ οι ασφαλέ, αλλά μπορεί να γίνει μια προφορική τροπολογία εδώ πέρα για το πεδίο εφαρμογή για να είναι ξεκάθαρο για τον καθένα πω τα ασφαλιστικά συμβόλαια δεν εμπίπτουν σε αυτήν εδώ την κατηγορία. Μετά. Μετά έχουμε άλλη μια τροπολογία του συναδελφού Πρεσέντο που λέει. Πώς να το εξηγήσω τώρα. το δικαίωμα το οποίο δίνουμε εδώ πέρα είναι ε, κάτι το προαιρετικό αλλά η τροπολογία του κυρίου Πρεσέδο λέει πως, πως πρέπει να εμποδίσουμε πως ε, θα αντικαταστήσουν τα κράτη-μέλη το δικό τους δίκαιο από αυτό εδώ πέρα. Μα δεν θα το κάνει κανένα κράτος μέλος να αλλάξει πλήρως το εθνικό του δίκαιο και να το κάνει ίδιο με αυτό εδώ πέρα το ευρωπαϊκό σύστημα. Εγώ λοιπόν αντιλαμβάνομαι την ε, τροπολογία Πρεσέδο ε, ότι θέλει να το κάνει αυτό πιο, πιο δύσκολο. Αλλά αυτό δεν είναι παρέμβαση στο εθνικό δίκαιο, δεν νομίζω. Πάει πολύ μακριά μετά. Μετά έχουμε τροπολογίες για τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Πάλι ε, τους Πρεσέδο για να εισαχθεί ένα είδος toolbox, όπως το λέει, για να γίνει το σύστημα αυτό κάπως πιο φιλικό προς το χρήστη. Σύμφωνα εδώ πέρα πλήρως, είμαι υπέρ και να έχουμε και υποδείγματα συμβάσεων. Πρέπει να είναι ξεκάθαρη σχέση μεταξύ διαφόρων νομικών μέσων πράγματι. Καλό αυτό, αλλά δεν ταιριάζει εδώ πέρα. Προσπαθήσω να το βάλω σε ένα άλλο άρθρο, σε ένα εκτιμώντας. Και βεβαίω μπορούμε να βάλουμε μια προφορική τροπολογία έτσι ώστε να περιέχει αυτό το toolbox ας πούμε κάποιες ε, επεξηγηματικές κατευθυντήριες γραμμές ε, για να ξέρει κανείς τι μπορεί να κάνει. Κατόπιν το έκτο σημείο ήταν αυτό και περνάμε στο παράρτημα που νομίζω αφορά γενικώ τις ε, συμφωνίες που βρισκόνται στη βάση όλων των ε, συστημάτων βεβαίως του δικαίου, αλλά θα πρέπει να αποτρέψουμε το να διαλέγει κανείς μόνο τα στοιχεία που τον ε, βολεύουν. Εδώ πέρα είναι η τροπολογία 21 του Σάντσες Πρεσέδο. Αλλά νομίζω πως δεν χρειάζεται αυτή η τροπολογία γιατί το να διαλέγει κανείς ούτως ή άλλως απαγορεύεται στο άρθρο 8 του τίτλου ας πούμε και της επικεφαλίδας και βεβαίως ε, αυτά είναι και στην ε, κατεύθυνση των σχέσεων B2C επιχειρήσεων με καταναλωτών οπότε ε, νομίζω πως μπορούμε να απλοποιήσουμε εδώ πέρα την κατάσταση. Οπότε δεν συμφωνώ με την τροπολογία σαν τις αλλά θα προσπαθήσουμε να το βάλουμε κάπου αλλού. Μετά έχω και ένα έβδομο σημείο. Η διαφορετική ερμηνεία που μπορεί να υπάρξει σε ζητήματα τα οποία δεν ρυθμίζονται. Έχουμε και πάλι τροπολογία του Σάντσες Πρεσέδο για να αφήσουμε την ερμηνεία στο εθνικό δίκαιο και όχι, όπως αναφέρει η πρόταση, να γίνεται η πρόταση, η ερμηνεία με συγχωρείτε με βάση τα ίδια τα εκτιμώντας της πρότασης. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει μία ενιαία ερμηνεία ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν πιο ενιαία. Δεν μπορούμε να λέμε πως θα έχουμε εθνικές ερμηνείες, θα έχουμε ένα μέσο με 27 διαφορετικές ερμηνείες. Δεν είναι αυτό εσωτερική αγορά αλλά μπορώ να κάνω μια πρόταση και να πούμε πως εκεί πέρα που υπάρχει αμφιβολία η νομική ανασφάλεια πρέπει τα κράτη-μέλη να ερμηνεύουν το δίκαιο στο μέτρο του δυνατού. Όπως λέει εδώ πέρα και στην αρχή της αυτή η πρόταση, εντάξει, γιατί θα υπάρχουν κενά και θα πρέπει να γεφυρωθούν κάπως. Οπότε, θα έλεγα πως πρέπει η ερμηνεία να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρωπαϊκή για να διαφυλάξουμε την εσωτερική αγορά. Για να διατηρήσουμε το σύστημα αυτό. Αλλά θα καταθέσω μια προφορική ε, τροπολογία. Τις δε προφορικές τροπολογίες θα τις συναντήσω με τους διάφορους ε, σκιώδους ηγητές για να είναι όσο το δυνατόν πιο απλούστεροι η λίστα της ε, ψηφοφορία για όλες τις ε, κοινοβουλευτικέ ομάδες. Αλλά νομίζω θα είναι ούτως ή άλλως απλά τα πράγματα. Δύο-τρία πραγματάκια ακόμα κύριε Πρόεδρε. Ε, επιπρόσθετη υποχρέωση για προσυμβατική ενημέρωση στα σημεία 23, 24, 25 και 26. Βεβαίω δεν μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα εκεί πέρα και αυτό αφορά νομοτεχνικούς λόγους. Όσον αφορά το 23, 24 και 25, αυτά αφορούν άρθρα του δικαίου των πολίσεων, τα οποία είναι κατά λέξη οι ίδιες προσυμβατικές υποχρεώσεις με αυτές που έχουμε στην οδηγία προστασίας των καταναλωτών, η οποία βεβαίως προσφέρει μια μέγιστη εναρμόνιση ενώ εδώ πέρα οι συνάδελφοι ξέρουν πως ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συζητήσεις οπότε εγώ θα έλεγα να μην το μπλέξουμε περαιτέρω το σύστημα. Υπάρχει τώρα η οδηγία οπότε εδώ πέρα είναι ταυτόσιμη η ορολογία που έχω υιοθετήσει και μετά έχουμε το σημείο 26 όπου υπάρχουν τροπολογίες και εδώ πέρα είναι το άρθρο 5 της Οδηγίας Προστασίας των Καταναλωτών. Εκεί πέρα υπάρχει μια ελάχιστη εναρμόνιση και νομίζω πως θα μπορέσουμε να βρούμε μαζί μια καλή τροπολογία. Αν δεν κάνω λάθος δε αυτή ήταν η τροπολογία του Sven Giegold. Και μετά, τέλος, κύριε Πρόεδρε είχαμε τροπολογίες που αφορούσαν καταχρηστικούς όρους και λέμε αν σε μια συμφωνία υπάρχουν ρήτες οι οποίες δεν επιτρέπεται τελικά να υπάρχουν, τότε η σύμβαση αυτή θα δεσμεύει για το κομμάτι το οποίο περιέχει ε, τους κανονικούς ε, όρους αλλά όχι για Δεν ξέρω εάν μπορούμε να θέσουμε ένα τέτοιο κανόνα γιατί εδώ πέρα αυτό το οποίο προτείνεται είναι ότι θα εκπληρώσει μόνο τους, θα εκπληρώσει υποχρεώσει του μόνο αυτός ο οποίος δεν έχει βάλει καταχρηστικούς όρους. Δεν έχει νόημα αυτό. Δηλαδή αν κάποιο έχει βάλει λάθος όρους συμβόλαιο, εγώ αγοράζω ένα ψυγείο, μου το φέρνουν που είναι το μέρος που έχει να εκπληρώσει ο πολιτή και εγώ δεν πληρώνω που είναι το μέρος που έχω να εκπληρώσω εγώ αγοραστής είναι κάπως υπερβολικό. Απλά νομίζω πως μπορούμε να αφήσουμε ένα κάπως ε, ένα αρκετά μεγάλο περιθώριο, αλλά όχι να είναι τόσο ριζική η τιμωρία. Τέλος πάντων θα τα δούμε αυτά με τους χειώδες ηγετές, αν μπορέσουμε να συμβιβαστούμε. Θα τα βάλουμε μετά ως ε, προφορικές ε, τροπολογίες για να βελτιώσουμε αυτή την γνωμοδότησή μας στην Νομική Επιτροπή, αλλά κυρίως είμαι γνώμων για το ότι ε, προσπαθούμε. Βεβαίως εμείς δεν είμαστε οι νομικοί, αυτή είναι η δουλειά της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων. Απλά είδαμε τα σημεία τα οποία είναι σημαντικά για εμάς. Οπότε νομίζω πως θα μπορέσουμε να καταθέσουμε κάποιες προφορικές τροπολογίες για να ξέρουν όλοι τι ε, ψηφίζουν για να είναι και ξεκάθαρος ο κατάλογος της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τάισεν. Πάμε στους κοιόδης εισηγητές. Ο κύριος Πρεσέδο. Έχετε το λόγο. Eh, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ θερμά και την εισηγήτρια για την ανάλυση που μας έκανε των τροπολογιών. Εγώ ε, υποβάλλω την ε, τη υπό το πρίσμα των, της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Δεν μιλούμε για το κόστος των, διαφορών. Μας ενδιαφέρουν το κόστος των συναλλαγών. Και η ποικιλομορφία, η διαφορετικότητα δεν είναι κατά ανάγκη κόστος αρνητικό, μπορεί να είναι αξία. Καλό θα ήταν όμως να έχουμε ένα κατόφλι προστασίας του καταναλωτή πιο υψηλό. Γιατί και σε επίπεδο συμβάσεων πρέπει να υπάρχει αρχή της ε, ελευθερίας των συμβάσεων. Η ποικιλία, η διαφορετικότητα είναι μία αξία, ένα πλεονέκτημα και το θέμα είναι να την ε, αξιοποιήσουμε με διπλό τρόπο. Αυτό το μηχανισμό μπορεί να μειώσει το κόστος των συναλλαγών. Στο μέτρο που στις διεθνείς ε, συναλλαγές θα έχουμε ένα αξιόπιστο μηχανισμό που θα μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης θα πρέπει να είναι προαιρετικό αυτό το σύστημα, να μην είναι ομοιόμορφο, ομοιογενές που να περιορίζει την ποικιλία, την ελευθερία τη, της συναλλαγής και την ελευθερία του καταναλωτή. Αυτό ο προαιρετικός χαρακτήρας είναι πολύ σημαντικός και από τη στιγμή που θα είναι προαιρετικό το σύστημα θα πρέπει να είναι στη διάθεση όσων το χρειάζονται αυτό το μηχανισμό. Δεν πρέπει να το περιορίσουμε σε συγκεκριμένη κατηγορία. Βέβαια, οι φυσικοί παραλήπτες είναι οι καταναλωτές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές ε, καταβάλουν το μεγαλύτερο κόστος συναλλαγής ε, σε περίπτωση που για κάθε συναλλαγή θα έπρεπε να έχουν ε, μία σύμβαση υπόδειγμα, ενώ οι πολυεθνικές εταιρείες ήδη δίνουν τα δικά τους υποδείγματα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που έχουν οι συναλλαγέ του. Να είναι λοιπόν προαιρετικό αυτό το σύστημα. Δεύτερον, να υπάρχει ένα προαιρετικό σύστημα που να συμβάλλει στον περιορισμό του κόστου, όπω λέω και εγώ στι ε, τροπολογίε. Όταν μιλώ για συμπληρωματικά εργαλεία, αυτό ακριβώ εννοούσα. Η συγκήτρια μίλησε για μια σύμβαση υπόδειγμα, μια στάνταρ σύμβαση. Στι αιτιολογικέ σκέψει, εγώ προσπάθησα ε, να συμπεριλάβω αυτή την ιδέα και στο διατακτικό, δηλαδή να έχουμε συμβάσει με τυποποιημένους όρους, ε, υποδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιούνται. Επίσης η αναθεώρηση θα πρέπει να ε, αξιολογεί και το επίπεδο αποδοχής. Επίσης αν μειώνει το κόστος συναλλαγής. Αυτό μας ενδιαφέρει για να αξιοποιηθεί από την οικονομία και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στους ευάλωτους καταναλωτές, δηλαδή στους πιο ευάλωτους χρήστες γιατί για αυτούς τους ευάλωτους χρήστες ε, χρειάζεται ένα τέτοιο εργαλείο, ένα τέτοιο μηχανισμό για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη τους. Επίσης, θα εξαιρέσουμε κάποιες διατάξεις ή όχι. Καταρχήν, να υιοθετήσουμε τη θετική αρχή, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι να πούν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις συμβάσει στο σύνολο ή ένα τμήμα τους. Και να είμαστε και ρεαλιστές. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε μια τυποποιημένη σύμβαση, σύμβαση υπόδειγμα, αυτό όμω δεν εμποδίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν ό,τι προσαρμόζεται στις δικές τους ανάγκες. Υπάρχει και το θέμα των εκκρεμών θεμάτων. Αυτή η σύμβαση υπόδειγμα έχει κάποια κενά. Βέβαια τα κενά μπορούμε να τα επιλύουμε με βάση τους ε, προσανατολισμούς και τις αρχές, αλλά ίσως δεν αρκεί αυτό. Όταν υπάρχει κενό, και αν για το κενό αυτό υπάρχουν εθνικοί κανόνες, καλύτερα να ισχύσουν αυτοί. Φυσικά, τηρώντας τις αρχές και αυτής της κοινοτική ρύθμισης. Τώρα, σε περίπτωση κενού θα πρέπει να εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο εχέγγυο για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Και θεωρώ ότι η συγγήτρια με το, την προθυμία που έδειξε και το πνεύμα συνεργασίας θα υποβάλει και κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε στη συμφωνία εν ώψη της ψηφοφορίας. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρεσέδο. Ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, δεν έχω καμία τροπολογία κατά θέση γιατί συμφωνούμε σε πολλά με την κυρία Τάισεν, αλλά να πω κάποια πραγματάκια. Δύο πράγματα γνωρίζουμε όλοι. Πρώτον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν εκμεταλλεύονται αρκετά την εσωτερική αγορά. Είτε γιατί χρησιμοποιούν και δεν μπορούν να εφαρμόσουν το εθνικό τους δίκαιο σε διεθνείς συναλλαγές, είτε γιατί βασίζονται σε Άλλε συμβάσει οι οποίε δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να αξιολογήσουν νομικά. Οπότε είναι μη ρεαλιστικό να υποθέσουμε πως ε, μπορεί κάποιος να αντικαταστήσει 27 διαφορετικά δίκαια των πολίσεων με ε, ένα ενιαίο ευρωπαϊκό. Οπότε έχουμε ένα προαιρετικό 28ο σύστημα, κάτι το οποίο είναι απολύτως θετικό Τώρα του έλωσε για την πρόταση να το αποστείλουμε πίσω, δεν έχει πολύ νόημα εμεί απλά μια γνωμοδότηση κάνουμε. Τώρα, για την ε, πρόταση και τροποποίησή της όπως προτείνουν διάφοροι συνάδελφοι για το εάν θα υιοθετηθεί στην πράξη, αν θα βοηθήσει στην πράξη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν την εσωτερική αγορά, αυτό θα το δείξει μόνο το μέλλον. Α, καλό να προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Και μετά από κάποιο καιρό, τώρα δύο, τέσσερα χρόνια, να επανεξετάσουμε τι έχει γίνει και βεβαίως αυτό δεν επιτρέπεται να οδηγήσει στο να προσθέσουμε ένα 28 σύστημα στα 27 ήδη ε, περίπλοκα και έτσι να δημιουργήσουμε μόνο περιπλοκές. Τώρα, εάν λειτουργήσει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για B2B, μεταξύ επιχειρήσεων δηλαδή, δεν θα το απέκλεια. Εάν γίνει μετά, όπως λέει ο Sven και σε άλλους τομείς, πρέπει να το δούμε τότε. Από τις διάφορες συζητήσεις που είχα εγώ με προσώπους ε, εμπορικών συλλόγων κτλ. Ε, εντάξει, είναι συγκρατημένα αισιόδοξη, θα έλεγα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πράξη με αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ κύριος Γκίγκολτ. Thanks, Chair. Ευχαριστώ. Ακόμη δεν έχω καταλάβει ποια ομάδα προηγείται. Αλλά φίλοι είμαστε δεν πειράζει. Πάντως, ε, καταρχήν δεν ε, προηγούμαστε εμείς. Στην Ολομέλεια ισχύει μάλλον αυτό. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και ευχαριστώ για τη θετική της αντίδραση σε ορισμένες τουλάχιστον τροπολογίες μας. Γενικώ συμφωνούμε με την πρόταση Επιτροπής πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τις ε, μικρές επιχειρήσεις και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ε, κοινή αγορά. Επίσης, ενστερνιζόμαστε την προσέγγιση της εισηγήτριας για τη διευκρίνηση του αποκλεισμού των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επίσης, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει κατάρτιση σε επιχειρηματίες, σε νομικούς και να ε, διευρύνει το πεδίο εφαρμογή σε κάποιες συμβατικέ συμφωνίες που δεν καλύπτονται από το κοινοτικό ευρωπαϊκό δίκαιο απολύσεων, αλλά επηρεάζονται από τα εθνικά νομικά πλαίσια, για παράδειγμα μεταβίβαση κυριότητας. Επίσης, έχουμε συντάξει κάποιες τροπολογίες. Θα επικεντρωθώ στα άρθρα μόνο. Στο άρθρο 6.2 μπορούμε να είναι συναφής η πληροφορία αυτή με την, με εξαίρεση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και οι συναφείς υπηρεσίες δεν καλύπτονται. Άρθρο 7, παράγραφος 1. Η προτινόμενη απαγόρευση της χρήσης ε, του κοινοτικού συστήματος πωλήσεων για συμβάσεις ε, μεταξύ εμπόρου που δεν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυθαίρετη. Προτιμούμε ε, το άρθρο 13, γιατί ο περιορισμός μπορεί να μην ε, ισχύει για διασυνοριακό εμπόριο. Προτείνω να είμαστε πιο σαφείς και μια και ζητούμε από τα μέρη να κάνουν το opt να υπαχθούν, προτείνουμε να καταργηθεί αυτός ο περιορισμός. Επίσης, διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ μεγάλων εταιριών ε, μπορεί να επωφεληθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πολίσεων. Τώρα, άρθρο 15 ε, σχόλιο συναφές με το προηγούμενο. Να προβλέψουμε την αναθεώρηση για, τις, ε, για την υπαγωγή των συμβάσεων ε, που δεν, που δεν συνάπτονται μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τώρα, σε ό,τι αφορά το παράρτημα κατά πόσο σε μία ανοιχτή σύμβαση μπορεί να αλλάξει η περιοδική τιμή, θα πρέπει οι καταναλωτέ να ενημερώνονται για προηγούμενε αλλαγέ των τιμών στα πλαίσια τη ε, συνολική ενημέρωση για τι τιμέ. Και όταν ε, το ποσό του λογαριασμού υπολογίζεται με βάση συναλλαγματικέ ισοτιμίε, θα πρέπει να προσδιορίζεται πώ προσδιορίζονται αυτέ οι συναλλαγματικέ ισοτιμίε. Και τέλο, αν υπογράφεται ε, το συμβόλαιο στην έδρα του εμπόρου, ή εξ αποστάσεως, άρθρο 25. Δεν ξέρουμε γιατί θα πρέπει ο καταναλωτής ε, να επωφελείται από την ενημέρωση για τις τιμές που προβλέπει το άρθρο 40. Ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν διστάμενες απόψεις για το θέμα αυτό και είναι κάπως περίεργο γιατί στην Επιτροπή ΙΜΚΟ σίγουρα η κρατούσα γνώμη είναι διαφορετική, διαφορετικές απόψεις. Το ίδιο εδώ επίσης η Νομική Επιτροπή έχει τη δική της άποψη. Υπάρχει λοιπόν διάσταση απόψεων, ακόμη και από ομοειδεάτες ή από, ε, από ευρωβουλευτές της ίδιας χώρας. Ανάλογα από το σε ποια επιτροπή ε, νίκει ο καθένας έχει και διαφορετική γνώμη. Συνήθως ομοειδεάτες έχουν την ε, ίδια γνώμη γιατί συνήθω όταν ομοδιώτε έχουν διαφορετική γνώμη, κάπου υπάρχει πρόβλημα, κάπου ίσω έγινε εσφαλμένη κρίση, υπήρξε λανθασμένη κρίση. Ίσως θα πρέπει οι εκπρόσωποι των ομάδων να συζητήσουν αυτό το θέμα, γιατί άνθρωποι που χαίρουν σε εμπιστοσύνη μου ε, συμφωνούν ότι αυτή η διαφωνία είναι προβληματική. Εμείς ε, ως ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ είμαστε υπέρ βέβαια αυτής της άποψης, αλλά καλύτερα να τη συζητήσουμε πιο διεξοδικά και να διευκρινίσουμε και την επιχειρηματολογία. Γιατί μπορεί η δική σας ομάδα να είναι κάπως πιο συνεκτική, αλλά στις άλλες ομάδες υπάρχει διχόνοια. Υπάρχουν τεράστιες εσωτερικές διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Και αυτό είναι που με προβληματίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σαΐντ Καμάλ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Χαίρομαι γιατί ο σοφός συνάδελφος των Πρασίνων μίλησε πριν από μένα. Ε, με εξυπηρετεί αυτό γιατί μου κάνει και πολύ καλή εισαγωγή για τη δική μου θέση. Άκουσα την εισηγητρία και τους σκιώδης εισηγητές και είναι ε, λογικό να πούμε ότι, κανείς, ε, ότι ε, μπορεί να αισθάνεται ότι διαφέρει πλήρως με τους, διαφωνεί πλήρως με τους προαναλύσαντε, αλλά αυτό δεν πρέπει να τον εμποδίζει να εκφέρει τη γνώμη του. Τώρα, ως προς τις αρχές, η νομοθεσία θα πρέπει να θεσπίζεται μόνο αν υπάρχει αποχρό λόγος για την ύπαρξή της. Και στην περίπτωση του κοινοτικού ευρωπαϊκού δικαίου δεν έχουμε πιστεί για κάτι τέτοιο, για την α, αναγκαιότητα μιας τέτοιας νομοθεσίας. Ο Σβέν έκανε μια πολύ καλή επισκόπηση και αξιολόγηση της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταξύ των ομάδων και μεταξύ των διαφόρων επιτροπών. Ε, αυτό που με προβληματίζει είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, γιατί πολύ συχνά ασχολούμαστε με οδηγίε και κανονισμούς και πολύ συχνά μπορούμε να προβλέψουμε την προσέγγιση του καθενό Άλλοι είναι υπέρ τη αγορά, υπέρ τη ρύθμιση, Στο συγκεκριμένο θέμα, με εντυπωσιάζει η συνένεση και από τις ε, από τους καταναλωτές, από τους επιχειρηματίες, ε, από τις κρατικές αρχές. Όλοι συμφωνούν ότι η πρόταση αυτή είναι περιττή και μπερδεύει τα πράγματα και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Κανένας δεν είπε ότι είναι καταπληκτική πρόταση και τη χρειαζόμαστε κατεπηγόντως. Δεν νομίζω ότι έχει πιστεί κανένας γιατί όπως είπε και ο κύριος Κλίντς δεν υπάρχει ενθουσιασμός, ε, αν μη τι άλλο. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, αλλά όλοι συμφωνούμε, έχουμε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλοι λατρεύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι αγαπημένες όλων και όλοι αισθανόμαστε ζεστασιά στην καρδιά όταν μιλούμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, δεν θέλει κανείς να πει τίποτα αρνητικό, αλλά ε, εγώ είμαι κατά της πρότασης αυτής. Δεν μ' αρέσει ε, να απορρίπτω ριζικά τα πράγματα, αλλά είμαι υπέρ του ρεαλισμού και προσπάθησαν κάποιοι συνάδελφοι με να βελτιώσω την πρόταση και βλέπω ότι όλες οι ομάδες προσπάθησαν και δεδομένου ότι είμαι σε αυτή την επιτροπή, μπορεί να είμαι εδώ μειοψηφία, μπορεί να είμαι και απομονωμένος και θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να εξετάσω σοβαρά όλες τις προτάσεις για να δω ποιες είναι οι πιο αξιόλογες. Και σίγουρα και οι σκιώδεις ηγητές από άλλες ομάδες υπέβαλαν πολύ λογικές προτάσεις. Πάντως η ΙΜΚΟ ζήτησε μελέτη επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο για την πρόταση και υπογράμμισε τις αδυναμίες της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό είναι το θέμα. Δεν ζητώ απόρριψη ελαφρά την καρδία. Είναι... Δεν είναι ότι θέλω να εξαφανιστεί τελείω αυτή η πρόταση, αλλά θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση που θα μπορέσουν να στερηθούν και οι καταναλωτές και οι επιχειρηματίες και οι νομομαθείς και οι κρατικές αρχές να συμφωνήσουν όλοι για το τι είδους κοινοτικό δίκαιο πωλήσεων θέλουν. Γιατί έχουμε διαφορετικές απόψεις και για το κατά πόσο χρειαζόμαστε ρυθμίσεις. Πάντως πιστεύω θα πρέπει να ξαναρχίσει το θέμα αυτό από την αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε σωστές διαβουλεύσεις και να συντάξει και μελέτη επιπτώσεων. Γιατί θέλουμε ομοιο... ενότητα και ομοιομορφία δεν θα προέλθει από τις διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων ομάδων και προστασίας καταναλωτών, αλλά από την υποστήριξη που θα δώσουν στην πρόταση. Ε, ξέρω ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν θα ήθελε να παρέμβει. Έχουμε καθυστερήσει κατά 10 λεπτά. Αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα με το χρόνο. Ήδη είχαμε πρόβλημα και το πρωί. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση θα ξαναδώσω λοιπόν το λόγο στην Μαριάν για να απαντήσει πολύ σύντομα παρακαλώ. Δεν θέλουμε να μας ξεφύγει ο χρόνος εδώ πέρα. Έχουμε και την ακρόαση. Σύντομη. Γιατί ξέρουμε όλοι νομίζω τι πρέπει να κάνουμε. Για αυτό το οποίο είπε τώρα ο συνάδελφος Κιμόβουλ. Αυτή την εβδομάδα οι συντονιστές στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα κάνουν μια προσπάθεια για να ζητήσουν από την ε, ομάδα αντικτύπου, μελέτης αντικτύπου του Κοινοβουλίου να δει το θέμα και έτσι Κομισιόν. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε και εμείς ε, την ε, πτυχή, όχι την ε, νομική, η οποία αφορά την Επιτροπή Νομικών ε, Θεμάτων, αλλά την ε, οικονομική, η οποία μας αφορά και βεβαίως να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα απλό σύστημα το οποίο θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν βεβαίως διάφορα προβλήματα, αλλά αυτά θα τα δει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, γιατί μετά ξεπερνάει τις δικές μας αρμοδιότητες, θα δουν εκεί πέρα οι αρμόδιοι νομικοί. Εμείς μπορούμε απλά να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας στην Επιτροπή αυτή και η Επιτροπή αυτή θα κάνει την αξιολόγηση αντικτύπου ξανά και θα μελετήσει τι μπορεί να γίνει και μετά ο καθένας στην ομάδα μας θα κάνει την επιλογή του για το τι θα γίνει στην ε, Ολομέλεια. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα νομίζω να αφιερώσουμε ε, περισσότερο χρόνο σε αυτό. Εμείς ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε στις 8 Οκτωβρίου. Δεν ξέρουμε πότε θα ψηφίσει η Επιτροπή η αρμόδια, αλλά δεδομένη τη βαριά ημερήσια διάταξη, ε, ε, καλό είναι να προχωρήσουμε το σύντομότερο δυνατόν. Σα ευχαριστώ λοιπόν, σα ευχαριστώ που ήσασταν όλοι σύντομοι και τώρα περνάμε στο σημείο 9, που είναι οι λειτουργίε διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κεντρικά αποθετήρια τίτλων και θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην Κέι Σουίνμπερν, για να μα παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσή. της. Παρακαλώ, Κέι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια στην Επιτροπή μα, αλλά και αλλού, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές της διαδικασίας συναλλαγή στις χρηματαγορές. Τη ε, της ε, την ε, διάσταση της συναλλαγή. Και αυτή τη στιγμή ένα συνάδελφο ε, στα πλαίσια αυτή τη επιτροπή δουλεύει ακόμα για να καλύψουμε όχι μόνο τι ε, μετοχέ, αλλά όλους, ε, όλες τις αξίες, κανόνες συμπεριφοράς, κανόνες για τι παρατυπίε και, τα κεντρικά, και κανόνες για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Υπάρχει τελευταία, η τελευταία ψηφία, που είναι η τελευταία φάση τη διαδικασία, που είναι ο διακανονισμός. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να το ρυθμίσουμε, με αυτό το κείμενο. Είναι ένα τεχνικό κείμενο βέβαια, παρόλα αυτά προσπάθησα να αξιολογήσω στην έκθεσή μου ε, όλο το μηχανισμό σαν να ήμουν ένας Ευρωπαίος ε, επενδυτής που θα υποφεληθεί από τη μείωση του κόστους, από την αυξημένη αποτελεσματικότητα στο σύστημα. Σε αυτή την πρόταση λοιπόν υπάρχουν δύο στόχοι. Καταρχάς η πρώτη έγινε πριν από πολλά χρόνια για τον κατακαιρματισμό ή μάλλον για την εξάλληψη των φραγμών στην ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τελικός στόχος να μειώσουμε το κόστος για τις διασυνοριακές συναλλαγές που αντιμετωπίζει ο τελικό επενδυτή. Από τη χρηματοπιστωτική κρίση έχουμε και έναν άλλο στόχο που είναι πολύ σημαντικό για όλου μα εδώ, αλλά και όχι μόνο εδώ. Θα πρέπει οι χρηματοταγορέ και οι υποδομέ των χρηματαγορών να είναι πιο σταθερέ και όπου μπορούμε να μειώσουμε το συστημικό κίνδυνο συνολικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Έχουμε 932 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ε, υπάρχουν πολλοί συμμετέχοντες ε, που συμμετέχουν στη διαδικασία διακανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ε, από κάθε άποψη υπάρχουν, είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία για τις υποδομές των χρηματογρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά υποστήριζω την πρόταση της Κομισιόν και τη γενική κατεύθυνση που έχει πάρει με την αρχική της έκθεση την οποία επεξεργαζόμαστε τώρα, στις τροπολογίες που υπέβαλα προσπάθησα να εστιάσω λιγάκι περισσότερο στην ενιαία αγορά και λίγο περισσότερο ε, στους στόχους που θέλουμε να υλοποιήσουμε για τις υποδομές των χρηματαγορών. Προσπάθησα να βάλω και ευελιξία όπου χρειάζεται, όπου γίνεται στην πρόταση της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο λοιπόν της, του διακανονισμού, πιστεύω ότι ο στόχος που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα αξιόγραφα που θέλει τυποποίηση του κύκλου διακανονισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να είναι αποτελεσματική η όλη διαδικασία, είναι σωστή. Παρότι κάποιες αγορές μπορούν να πάνε πιο γρήγορα από το τι του, είναι σημαντικό να έχουμε ένα νούμερο αρχικά ε, και αυτό είναι ο στόχο μα. Το τι του νομίζω ότι είναι ο λογικός τρόπος ε, να ξεκινήσουμε, αλλά θα πρέπει μακροπρόθεσμα να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουμε αυτό το στόχο, τι 2. Αλλά μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε μια αναθεώρηση, να φτάσουμε στο T plus 1 ή και κάτω. Ε, φυσικά, όσο μικρότερη περίοδος ε, αβεβαιότητας ανάμεσα στους δύο συναλλασσόμενους, τόσο καλύτερα για το σύστημα. Θέλω να υπάρχουν καλοί κανόνες για το διακανονισμό και υποστήριζω την πρόταση της Κομισιόν για ε, κυρώσεις, ούτως ώστε να, είναι, να γίνεται εμπρόθεσμα ο διακανονισμό, αλλά είμαι λίγο πιο προσεκτική. Μια και όλο το καθεστώ του διακανονισμού που προβλέπει η Κομισιόν, ε, έχει ένα υποχρεωτικό, εμπεριέχει ένα υποχρεωτικό καθεστώς αγοράς. Θέλω μεγαλύτερη ευελιξία ε, για κάποια προϊόντα, αυτά που είναι λιγότερο α πούμε ρευστά. Επομένω, στι τροπολογίε μου ε, λέω ότι με βάση τις στατιστικές ε, θέλω να πω ότι η αποτυχία η αδυναμία διακανονισμού συμβαίνει αρκετά, ε, υπά... εμφανίζεται ας πούμε, αλλά τελικά ε, επιλύεται μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θέλω λοιπόν η ακαμψία που προτείνεται να μειωθεί. Ειδικά, μια και το, αυτό το καθεστώς αγοράς ε, γίνεται αφού το ζητήσει ο αποδέκτης. Ξεκινάει αυτός δηλαδή την διαδικασία όταν θεωρεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχουμε τώρα ένα πολύ περίπλοκο σύστημα με διαφορετικά προϊόντα κτλ. Ε, δεν νομίζω ότι θέλουμε ότι είναι προς όφελος κανενός αυτό. Ε, θα πρέπει να το απλουστεύσουμε γιατί ε, ο τελικός αποδέκτης ούτως ή άλλως μπορεί να ζητήσει τη διαδικασία αγοράς. Ε, μια και όλοι έχουμε στο μυαλό μας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρθηκε ο συνάδελφος έτσι με τρυφερά λόγια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τους κανόνες για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν θέλουμε να εθαρρύνουμε ε, την ε, εισδοχή των ε, εταιριών αυτών στο χρηματιστήριο και την πρόσβασή τους στι στις ε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είναι ειδική κατηγορία και στα πλαίσια της MIFID. Θα λοιπόν στα πλαίσια αυτού του κειμένου να αναγνωρίσουμε αυτήν την ειδική κατηγορία και να βάλουμε κάποια ευελιξία ε, σε αυτό το τομέα που είναι λιγότερο ρευστό. Υπάρχει ένα παράθυρο 15 ημερών, όπου ε, τα μέτρα ε, του διακανονισμού δεν αρχίζουν να ισχύουν. Περιμένουμε 15 μέρε και μετά αρχίζουν να ισχύουν λοιπόν. Ούτω ώστε να μην εμποδίζουμε του επενδυτέ από τον συμμετάσχουν λοιπόν. Αυτή τη στιγμή Είναι σημαντικό να μάθουμε από τις εμπειρίες των ε, ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ε, προσπαθήσει να εισαχθούν στο σύστημα. Αν λοιπόν οι εταιρείε αυτές μπορούν να τα καταφέρουν μέσα στο διάστημα T συν 2, οκ. Okay. Αν όχι, λίγο μεγαλύτερη ευελιξία θα ήταν κακό. Τώρα, για... αποφάσισα ότι τα, ΚΑ, τα ΚΑΤ αυτή τη στιγμή λειτουργούν σε εθνική βάση τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Ε, νομίζω ότι έχει νόημα η, ΕΣΜΑ να κάνει μία αξιολόγηση. Γιατί ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι επαυξάνουν το συστημικό κίνδυνο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα απλής ε, κοινοποίησης. Ενώ όταν υπάρχει ε, μεταβίβαση του κινδύνου ε, στα πλαίσια του ΚΑΤ, τότε θέλω μεγαλύτερη αυστηρότητα. Ε, ο διακανονισμός δεν θεωρείται από τους επενδυτές ως το επικίνδυνο τμήμα της συναλλαγής. Εγώ ασχολήθηκα πολύ με θέματα προστασίας ε, των επενδυτών και στην ήθιτ και σε αυτή την πρόταση. Αλλά διάφορες μεγάλες εταιρείες που κατέρευσαν ανάγκασαν τους επενδυτές να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή, να γνωρίζουν που βρίσκονται τα, τα ταξιόγραφά τους, ε, τα περιουσιακά του στοιχεία κτλ. Επομένως υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα με, με το διαχωρισμό. Καλό είναι να ξέρουν που βρίσκονται τα περιουσιακά του στοιχεία και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ε, ανάλογα με το που βρίσκονται αυτά τα, σε ποια δικαιοδοσία ανήκουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται και τα νομικά του δικαιώματα και να μπορεί να έχουν πρόσβαση και στους ε, κινητές αξίες των συντομότερων δυνατών, στα αξιόγραφα των συντομότερων δυνατών. Έχω μπει και σε εδάφη που δεν έχει δίσδυση κομισιών. υπάρχουν θέματα εσωτερικοποίησης του διακαονισμού και επανυποθήκευσης. Είναι δύο όροι οι οποίοι δεν είναι πολύ... δεν Με βάση την έρευνα που έχω κάνει, ήταν δύσκολο να βρω πληροφορίε για αυτά τα δύο θέματα, γιατί τα δεδομένα δεν έχουν συλλεχθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά υπάρχει κίνδυνος ε, να... για όλο το σύστημα διακαονισμού με αυτά τα δύο ζητήματα. Οι δραστηριότητες της εσωτερήκευσης και της επανυποθήκευσης θα πρέπει να παρακολουθούνται και να υπάρχουν εκθέσεις προς, τους, ε, προς τις αρχές. Θα πρέπει να έχουμε στοιχεία για να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, ούτως ώστε στο μέλλον να είμαστε σε θέση να θεωρήσουμε τη διαδικασία, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι καλύπτουμε κάθε πτυχή και ότι δεν έχουμε δημιουργήσει ε, νέο παραθυράκι το, από το οποίο μπορεί να διαφύγουν διάφοροι. Επίσης, η, η Κομισιόν ζητάει τα ΚΑΤ ε, να λάβουν υπόψη τους τις τραπεζικές υπηρεσίες. Λύσεις ενίας αγοράς ε, είναι προτιμότερες από τις τα εθνικά opt-out ή από τις παρεκκλήσεις. Αν συνδυάσουμε τα ΚΑΤ και τα τραπεζικά, ε, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα συστημικού κινδύνου. Ίσως ε, θα ήταν καλύτερο να βρούμε μια άλλη λύση, χωρίς παρεκκλήσεις δηλαδή. Όπως είπα και στην έκθεσή μου, υπάρχει μια έκθεση της BIS για τους κινδύνους ρευστότητας. Στο, για το ΚΑΤ ε, βασιζόμαστε σε λίγες επενδυτικές τράπεζες ε, που θα δώσουν ρευστότητα και τι θα γίνει όταν εξαλειφθεί αυτή η ρευστότητα, δεν υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Τι θα γίνει αν μία από αυτές τις τράπεζες σταματάει την παροχή ρευστού για εμπορικούς λόγους. Νομίζω ότι υπάρχει ένα συστημικό θέμα εδώ, κινδύνου δηλαδή, που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ε, δεν νομίζω ότι με τι δύο νομικέ οντότητε επιλύεται το πρόβλημα, όπω λέει η Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια νέα τράπεζα διακανονισμού σε περίπτωση κρίση που θα λύει το θέμα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη των σχεδόν εισηγητών και των άλλων μελών τη Επιτροπή να μου πούν τι απόψει του για να δούμε πώ μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα στην ενιαία αγορά. Νομίζω ότι πρέπει να ψάξουμε το θέμα πολύ προσεκτικά, το ρόλο του CISD, ε, γιατί Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα. Το, ο διακανονισμός είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας συναλλαγής και θα πρέπει να τους εξασφαλίζει απόλυτη ασφάλεια. Όλοι οι συμμετέχοντες αγοράς θα πρέπει να βρούμε λύσεις ενιαίας αγοράς για τις υπηρεσίες αυτές, να έχουμε ε, σταθερότητα, ανθεκτικότητα ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε όμως να φέρουμε και τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και φυσικά θα πρέπει να έχουμε νομοθεσία η οποία αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα και να αντιμετωπίζει και τα προβλήματα καθώς τα εμφανίζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τους σκιώδης ε, και αν θέλει κάποιος άλλος να λάβει μέρος στη συζήτηση, παρακαλώ να, τον δηλώσει, να το δηλώσει πέραν των σκιωδών εισηγητών για να δω πόσο χρόνο θα δώσω στον καθένα. Εκ μέρους του ΕΛΚ, ο Χέρπερτ Ντόρφμαν. Ευχαριστώ. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κέι Σουινμπορν μετά τις συζητήσεις που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες και για τα πολλά ζητήματα που ανέφερε με τα οποία συμφωνώ πλήρως. Αλλά νομίζω πως δύο ζητήματα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η ασφάλεια και η εσωτερική αγορά. Περισσότερη ασφάλεια και περισσότερη εσωτερική αγορά. Περισσότερη εσωτερική αγορά εδώ πέρα σημαίνει περισσότερος ανταγωνισμός σε μια αγορά η οποία de facto είναι πόλιο, γιατί υπάρχουν εθνικά κεντρικά αποθετήρια και σε ελάχιστο μισή υπάρχει εσωτερική αγορά. Οπότε νομίζω πως η πρόταση της Κομισιόν εδώ πέρα για εισαγωγή περισσότερο ανταγωνισμό είναι θετική. Θα ήθελα τώρα να αφαιρθώ σε ορισμένα σημεία από αυτά τα οποία είπε και η Σουίνμπορν. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε για κύκλους ε, απολογισμού. Η συγκίτρια είναι σωστό και αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν, αλλά νομίζω πως είναι λογικότερο να προβλέψουμε μεγαλύτερα διαστήματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα ήταν καλό να δημιουργηθεί μια ρύθμιση η οποία κάνει δύσκολη τη ζωή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το θέμα της επιτήρησης, επίβλεψης, δύο πράγματα θεωρώ πως είναι λογικό να σκεφτούμε μήπως η πρόταση της ε, Κομισιόν όσον αφορά την σύνδεση των ε, ΚΑΤ πηγαίνει πάρα πολύ μακριά και είναι πολύ γραφειοκρατική. Δεν είναι ανάγκη να υπάρξει πλήρης ε, τυποποίηση. Νομίζω πως μια ειδοποίηση για τη σύνδεση αυτή υπάρχει χωρίς να υπάρχει μια εξάντε αδειοδότηση. Επίσης δεν είναι να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Νομίζω δεν πρέπει να γίνει κατεύθυνση γιατί έτσι θα φερνάρουμε την εσωτερική αγορά. Και επίσης εδώ πέρα συμφωνώ με την Κέι Σούμπερν ε, για το ότι θα θέλαμε να μάθουμε τι προτείνει η Κομισιόν για την αδειοδότηση των ε, ΚΑΤ. Νομίζω πως αυτά είναι πολύ ουσιαστικές ε, απαιτήσει. Το βασικό θέμα και το πιο πολιτικό θέμα στην όλη υπόθεση είναι σε ποιο βαθμό πρέπει να έχουν άδειε τραπεζών τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Πέντε τέτοια στην Ευρώπη έχουν άδεια τράπεζας και δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στην εσωτερική αγορά και άρα διασυνοριακά και έτσι υπάρχει ίσως η αναγκαιότητα να διεξάγουν κάποιες τραπεζικές εργασίες, να έχουν κάποια χρήματα στη διάθεσή τους και αυξάνεται αυτή η τάση. Η Κομισιόν προτείνει μια εξαίρεση, μια ειδική ρύθμιση Εγώ θεωρώ πως πρέπει να βρούμε μια ρύθμιση που θα δημιουργήσει όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των κεντρικών αποθετηρίων. Και πρέπει να σκεφτούμε αν αυτή η εξαίρεση πραγματικά είναι η καλύτερη ή όχι ή μήπως θα ήταν καλύτερο να, επιτρέπουν, να επιτρέπουμε να κάνουν κάποιες τραπεζικές εργασίες σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Αυτό το οποίο βλέπω επιφυλακτικά είναι σε ποιο βαθμό οι λοιποί συμμετέχοντες στην αγορά, μη κεντρικά αποκτήρια δηλαδή, μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτών. Η Κομισιόν λέει πως πρέπει αυτή η δραστηριότητα να την κάνουν και αποκλειστικά κεντρικά αποκτήρια τίτλων και όχι τράπεζε και λοιποί συμμετέχοντες στην αγορά. Θεωρώ πως αυτά τα πράγματα σχετίζονται άμεσα γιατί Εάν απαγορεύουμε στα αποθήρια τίτλων να έχουν τραπεζικές άδειες, δεν μπορούν να είναι τράπεζες. Αντιστρόφως, εάν στις τράπεζες επιτρέψουμε να είναι κεντρικά αποθήρια τίτλων, ε, δημιουργούμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι και, και δίκαιη. Και έτσι αποδυναμώνονται ή τα υφιστάμενα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Και νομίζω και από πλευράς ασφάλειας και ελέγχου του διακανονισμού αξιογράφων δεν θα ήταν σωστό. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε το θέμα και θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια κατάσταση η οποία θα δημιουργεί ε, ίδιους κανόνες για την ίδια δραστηριότητα. Και τελειώνω με το εξής. Η συγκήτρια τόνισε πολύ περισσότερο τον ρόλο της ΕΣΜΑ, πολύ περισσότερο από την Κομισιόν και είναι λογικό αυτό. Αφού δημιουργήσαμε την ΕΣΜΑ πρέπει να της δώσουμε και τα ανάλογα καθήκοντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο είναι εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση που μας παρουσίασε, πραγματικά είναι διεξοδική, τεκμηριωμένη, προσέλκυσε πληθώρα τροπολογιών που άπτονται των πιο κεντρικών σημείων και έχει μια προσέγγιση για την εσωτερική αγορά που με βρίσκει σύμφωνο. Πρόκειται για πολύ σημαντικούς μηχανισμούς ε, για την ενίσχυση εμπιστοσύνης, ε, για τις διασυνοριακές συναλλαγές, όχι μόνο για τους επενδυτές που είναι αντισυμβαλόμενοι, αλλά και ως προς την ανάγκη να έχουμε πραγματικά αγορές ε, τίτλων που θα είναι διαφανείς, ασφαλείς είναι σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Επίσης έχουμε ένα μητρό τίτλων και για τη μεταβίβαση των τίτλων. Σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας μιας τέτοιας αγοράς. Και ένα άλλο σημαντικό είναι οι απαιτήσει ασφαλείας που αφορούν την νομισματική πολιτική και επίσης έχουν μεγάλη σημασία δεν αρκούν ε, οι συμφωνίες ε, των ε, αντισυμβαλωμένων. Χρειαζόμαστε μια κοινοτική νομοθεσία. Βέβαια ο κανονισμός δεν καλύπτει όλα τα σημεία, απαιτεί δύο από τις τρεις βασικές υπηρεσίες. Επίσης, σε ό,τι αφορά το target 2 securities και το ορίζοντας το 2015 δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια εκεί. Πολλά θέματα αναφέρονται. Το θέμα της τραπεζικής ε, άδειας, άδεια για τραπεζικές ε, εργασίες, γιατί θέλουμε να είναι περιορισμένη αυτή η άδεια για τις τραπεζικές εργασίες, αφενός και αφετέρου να αποσαφηνίσουμε το γεγονό ότι έχει κάποιο τέτοια άδεια, δεν σημαίνει ότι ήδη πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ε, για τέτοιο φορέα προϋποθέσεις που προβλέπει ο κανονισμός. Ένα σημαντικό θέμα είναι η αποϊλοποίηση των μετοχών. Ε, είναι, έχουμε κάποια ισοδύναμα, ισοδύναμους μηχανισμούς και αν υπάρχει διαφοροποίηση, διαχωρισμός ανάλογα με τους διάφορους φορείς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ίση μεταχείριση για ίσες δραστηριότητες. Η αρχή αυτή είναι σωστή και αυτή θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ίση πρόσβαση διαφάνεια για τους συμβαλόμενους, αλλά διαφάνεια και της αγοράς για τις διάφορες συναλλαγές που γίνονται. Θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, ταχεία, συναλλαγέ ε, συναλλαγές με χαμηλό κόστος, με ελαστικότητα, αναλογικότητα και μείωση των κινδύνων. Και φυσικά την απαραίτητη ασφάλεια με παροχή εγγυήσεων για τους πελάτες για τους δικαιούχους και γενικώ για τους φορείς αγοράς, αποφεύγοντας τη σύγκρουση συμφερόντων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για ε, ε φορείς που υποχρεούνται να εφαρμόσουν μια πειθαρχία και την αρχή της προφύλαξης και φυσικά να υπάρχουν κάποιες νέες απαιτήσει για τους διακανονισμούς η απόρριψη του εκδότη να είναι εξαιρετική περίπτωση, γιατί πρόκειται για σημαντικές υποδομές ε, της αγοράς. Επίσης, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται εξαιρέσεις για, τους, ε, για, ε, για την εκτέλεση των διαταγών. προτιμούμε ε, άδειες και όχι κοινοποίησεις και το θέμα της ισοδυναμίας θα πρέπει επίσης να στηρίζεται σε μια αρχή αμοιβαιότητας. Η αρχή της αμοιβαιότητας όταν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, εξασφαλίζει την ισοδυναμία. Για όλα αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, θα εκπονήσουμε κάποιες τροπολογίες. Πάντως η πρώτη μου θερμό αντίδραση μετά την παρουσίαση της ηγήτριας ήταν πολύ θετική και γι' αυτό τη συγχαίρω για το διεξοδικό και αξιόλογο έργο της που θα είναι πολύ χρήσιμο και θα αποτελέσει τη βάση για την υποβολή και των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η σκιώδη συγγήτρια για την ομάδα των φιλελευθέρων. Θα κάνω και εγώ ένα σχολιασμό. Ευχαριστώ, Κέι, γιατί με την έκθεσή σου που είναι πολύ μεστή και τεκμηριωμένη, μας διευκόλυνες και μερικές τροπολογίες τις έχεις, καταθέσει, τις καταθέσει ήδη, οπότε μας απαλλάσσεις από τον κόπο. Βέβαια, σε ορισμένα σημεία θα καταθέσω τροπολογίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει θέλω να σε υπονομεύσω, ούτε ότι η σιωπή μου είναι υποπτή. Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές άδειες, ένα θέμα που ανέκυψε. Πολύ σωστά είπες ότι ίσως εκεί υπάρχει δυνατότητα συστημικού συνδυασμού. Θα πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, γιατί όντως εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός και συμφωνώ ότι η διαγραφή της ε, εξαίρεσης είναι σωστή. Τώρα, αν δεν συμφωνήσουμε να διαγραφεί η εξαίρεση, τότε θα πρέπει τουλάχιστον να προσδιορίσουμε ποιες τραπεζικές υπηρεσίες καλύπτονται από τον διακανονισμό, αυτό το νομοθετικό αυτό κείμενο το τέταρτο νομοθετικό κείμενο για τους διακανονισμούς. Να ξέρουμε ποιες είναι οι απαιτήσει και επίσης να συνδέσουμε αυτό το θέμα με την, το θέμα της διευθέτησης της αντιμετώπισης των κρίσεων. Για να μην ε, λόγω του αδιέρετου χάσουμε και τις δύο πλευρές συμφωνώ να διαγράψουμε την εξαίρεση, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε, δεν συμφωνήσουμε, θα πρέπει τουλάχιστον να διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση που ισχύσει κάποια εξαίρεση, ε, να μην γίνεται ανεφόρον, να συνοδευτεί αυτή από κάποια αιρεσιμότητα και μάλιστα από πολύ αυστηρούς όρους που θα προσδιορίζονται και στα πλαίσια της ε, διαχείρισης των κρίσεων. Σε ό,τι αφορά την εσωτερήκευση, χαίρομαι που το ανέφερες. Δεν ξέρω αν αρκεί όμως η ετήσια έκθεση. Και από τη στιγμή που θα αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα θα πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο για την πρώτη ετήσια έκθεση. Καλό δεν είναι να υπάρχει μια ενδιάμεση ενημέρωση. Ίσως ε, τρίμηνη, γιατί όταν αρχίσει το target του security φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα περιμένει πιο τακτική ενημέρωση για να μπορούμε να παρακολουθούμε την αύξηση με την εφαρμογή του target του security. Βέβαια, από την άλλη θέλουμε να κάνουμε πολύ επαχθή τη διαδικασία. Να το συζητήσουμε όμως, να σκεφτούμε τι είδους τακτικότητα είναι απαραίτητη. Σε ό,τι αφορά τα ισοδύναμα, εδώ υπάρχει μια πληθώρα απόψεων και εγώ έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Ναι, μεν, ε, συμφωνώ ότι για τρίτες χώρες όλα θα πρέπει να είναι με βάση το αποτέλεσμα, γιατί αν, έχουμε, αν μία λυσίδα και την κόψουμε, δεν έχει σημασία πού θα κόπει. Το θέμα είναι να υπάρχει αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά τη νομική ισχύ των διαφόρων ρυθμίσεων για να μην ε, έχουμε πλήρη άγνοια για το τι ισχύει στο άλλο κράτος, στο τρίτο κράτος. Σε ό,τι αφορά το ΕΜΙΡ ε, και το ΜΙΦΙΤ, θα πρέπει επίσης να υπάρχει συνάφεια με τα δύο αυτά νομοθετήματα. Για το buy-in, συμφωνώ με την πρότασή σου. Δεν ξέρω, μήπως θα μπορούσαμε να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί και αντί να ε, να στηριχτούμε σε έναν ε, ορισμό της ρευστότητα, από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες ε, ε, περιπτώσεις που δεν υπάρχει ρευστότητα, αυτές να τις ορίσουμε. Ιδιαίτερα όταν αφορά αγορά μικρής κλίμακας ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί εκεί ίσως δημιουργηθούν διαταραχές. Γιατί περιμένουμε τον κανονισμό για τις ανοιχτές πωλήσει. Να μην επιδεινώσουμε δηλαδή την κατάσταση. Να δούμε τι θα γίνει και με εκείνο τον κανονισμό. Τώρα, αν ανακύψει το θέμα λόγω του μεγέθους της αγοράς, ε, να μην ε, τις πλήξουμε. Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν κάτι άλλο εδώ να επινοήσουμε σε περίπτωση της έλλειψης αυτής της ρευστότητας. Και τέλος, μια και τα υπόλοιπα σημεία καλύφθηκαν, είναι το θέμα της αποϊλοποίησης. Είπες ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη και την Ήδη τη μέρα της συναλλαγής. Δεν ξέρω όμως. Θα μπορούσαμε έτσι να μείνουμε στο πρότυπο της συνδύο. Θεωρητικά συμφωνώ ότι αυτός που έχει τη μετοχή έρχεται και μπορεί να την πουλήσει αυθημερών τη μετοχή, τον τίτλο. Αλλά αν δημιουργηθεί μια καθυστέρηση τότε το χρονικό διάστημα δεν μας ικανοποιεί παρακαλώ, ας και αυτό υπόψη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε εδώ μια μεταβατική περίοδο. Να πούμε ίσως αυθημερών, αλλά να μπορεί να είναι και πριν την συναλλαγή. Αυτά γενικώ πάντως συμφωνώ με τις προτάσεις σου και μπορούμε να ακούσουμε τον επόμενο σκιώδη συγητή από τους πράσινους, τον Σβέν. Uh, uh, Ευχαριστώ, Κέι, για την έκθεσή σου. Συμφωνούμε με πολλά από αυτά που είπες και έκανες. Και πριν μπω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας πω ότι πιστεύω ότι πρέπει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς το κόστος συναλλαγής στην Ευρώπη. Είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι ε, συμβαίνει στις Ηνωμένε Πολιτείε με το δικό τους επιχειρηματικό μοντέλο. Φυσικά εμεί έχουμε ξεκινήσει από αλλού. Αλλά τελικά ο στόχος θα πρέπει να είναι να μειωθεί αυτό το κόστος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να το επιτηρούμε εκ του σύνεγγυς αυτό το θέμα. Γιατί η αύξηση του κόστου συναλλαγή δεν είναι κοινωνικά υποφελής. Φυσικά είμαστε σε μια διαδικασία υπέρβασης κάποιων ιστορικών φραγμών που ακόμα και σήμερα κατακαιρματίζουν αυτή την αγορά. Και φυσικά δεν πρόκειται εν μία νυχτή να μειωθεί το κόστος συναλλαγής, αλλά πρέπει να μειωθεί. Τώρα μπαίνω στις λεπτομέρειες. Χαιρόμαστε με την ε, κατέθεση της πρότασης της Κομισιόν για τις τροπολογίες. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τις αγορές όπου συμμετέχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης ε, πιστεύω ότι τα ΚΑΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και είμαστε υπέρ των ε, σχετικών αλλαγών στο ε, εκτιμώντας 16 άρθρο και άρθρο 39 για την καταπολέμηση της απάτης. Είναι καλό να ευθυγραμμίσουμε τους ορισμούς με την οδηγία MIFID στο άρθρο 2 και επίσης μας αρέσει η ιδέα της τυποποίησης των τυποποιημένων εκθέσεων πληροφόρηση στο 6 α Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε και το άρθρο 7.1. Ετήσια έκθεση στατιστικών ε, λεπτομερών ε, για αποτυχία διακανονισμού. Ε, επίσης, στην αναθεώρηση από την έσμα του, των ΚΑΤ και στον τίτλο 2 και στο κεφάλαιο 3α, καλό είναι να εντοπίσουμε ε, την ε, εξωτερήκευση του διακανονισμού. Ε, γιατί υπάρχει και ένα τμήμα του διακανονισμού που δεν περνάει μέσα από τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Ε, υπάρχει περίπτωση εξωτερήκευσης αυτού του διακανονισμού, ε, ούτως ώστε μόνο οι εγκεκριμένοι, τα εγκεκριμένα αποθετήρια να μπορούν να προβαίνουν σε αυτόν τον διακανονισμό. Στο άρθρο 13.1 και στο άρθρο 23 συμφωνούμε με υποχρεωτικές επιθεωρήσεις, τουλάχιστον ε, ετησίως των προβληματικών κάτω. Στο άρθρο 31.6 συμφωνούμε με την πληροφόρηση που θα πρέπει να γίνεται προς τους χρήστες για τις υπηρεσίες των ΚΑΤ και στο 57 4ε λέτε ότι τα ΚΑΤ θα πρέπει να αντέχουν σε περίπτωση που μειωθεί η ρευστότητα από τους διάφορους παρόχους. Είναι σημαντικό για την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επίσης λέτε τα ΚΑΤ θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ε, ταυτόχρονη πτώχευση ε, άνω του ενός συμμετεχόντων. Εμείς θα λέγαμε να βάλετε κατευθείαν τουλάχιστον δύο. Στο 44.2 ζητάτε ε, το δικαίωμα των υποπτικών αρχών να ζητήσουν ε, αλλαγές στα σχέδια ανάκτησης ε, που έχουν τα ΚΑΤ. Και στο 52.2 λέτε να μην υπάρχει δυνατότητα κατά ανάγκη της εθνικής επιλογής για τα ΚΑΤ. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για τέσσερα σημεία. σε διάφορα άρθρα προτείνεται για το θέμα του διακανονισμού των αξιογράφων προτιμούμε την πρόταση της Κομισιόν που εγκρίνει μόνο τους, που επιτρέπει μόνο στα εγκεκριμένα ΚΑΤ να προβαίνουν σε αυτό το διακανονισμό. Η ανησυχία σου για την αλλαγή των πρακτικών μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις κατάλληλες διατάξεις, ούτως ώστε να δώσουν το χρόνο στα ΚΑΤ να αναδιοργανωθούν, ούτω ώστε να πάρουν και αυτή την έγκριση. Δηλαδή τα ΚΑΤ που δεν έχουν την έγκριση να την πάρουν. Για το 44α, το νέο. Να βάλουμε αυτόν τον περιορισμό για τη συλλογή των φόρων και να το βάλουμε αυτό στην, στις ιδέες μας. Είναι χρήσιμες πληροφορίες και νομίζω ότι το κράτος θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες. Έχουμε αρκετά προβλήματα ήδη με τη συλλογή των φόρων Πολλές φορές έχει πει το Κοινοβούλιο ότι χρειάζεται ε, και ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αν έχουμε τέτοια, τέτοιους φορείς, τότε δεν καταλαβαίνω γιατί το κράτος θα πρέπει να αποδυναμωθεί και να μην μπορεί να χρησιμοποιεί αυτές τις προφορίες. Το 7-2. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να κάνουμε αυτόν τον αποκλεισμό σε περίπτωση που υπάρχει καθυστερημένο ε, καθυστερημένος διακανονισμός. Ποιο ο λόγο που σα οδήγησε σε αυτό και στο 15, στο εκτιμώντας 15, διρωτόμαστε γιατί θα πρέπει η αγορά να ξεκινήσει μόνο σε περίπτωση που τη ζητήσει ο αποδέκτη. Δεν θα πρέπει να είναι αυτόματη διαδικασία ούτω ώστε να υπάρχει και προβλεψιμότητα και σταθερότητα τη διαδικασία του διακανονισμού. Όπω πάντα Κέι, με μεγάλη χαρά συνεργαστήκα μαζί σου. Περιμένουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι θα βρούμε μια καλή λύση. Ευχαριστώ και για την καλή αρχή και περιμένουμε να συνεργαστούμε μαζί σου και με τους άλλους συναδέλφους για την έκθεση. E, Γιώργεν από την ΚΟΕ. E. Ναι, ευχαριστώ. Από την ΚΟΕ e δεν έχουμε παρατηρήσεις αυτή τη στιγμή. Ζητώ συγγνώμη, θα τα πούμε στις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ένας άλλος. Όχι, οπότε επιστρέφουμε σε σένα, Και... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Νομίζω πως τα καλά είναι, είναι πως έχουμε μια συνένεση θα έλεγα σε ένα τεχνικό θέμα και είμαι σίγουρος πως οι υπόλοιποι θα προσπαθούν να αντιληφθούν το πολύ δύσκολο και στέγνο αυτό θέμα. Ελπίζω λοιπόν να μην είμαι μόνιμο και Βέβαια, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Υπάρχουν και πολλοί τομείς ε, ε, του οποίου βλέπω τώρα ξανά μετά το καλοκαίρι ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και βεβαίω αναμένω τη συνεργασία με τους κοιόδη ηγητέ για να μπορέσουμε να κάνουμε το κείμενο καλύτερο για την κοινή αγορά και να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι χωρίς πολλές ε, διαφωνίες ελπίζω. Ευχαριστώ. Ωραία ωραιότατα. Ξανακερδίσαμε τα δέκα μας λεπτά. Μήπως να ξανακάνουμε άλλο ένα γύρο. Όχι, όχι, εντάξει. Ξέρω πως έχουν έρθει οι άνθρωποι και περιμένουν. Η προθεσμία για τις τροπολογίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι η 18η Οκτωβρίου, εξέταση τροπολογιών 28 Νοεμβρίου. Θα ψήσουμε στην Επιτροπή 18 Δεκεμβρίου και θα πάμε στην Ολομέλεια. Πολλά πράγματα βλέπω. Τον Μάιο του 2013 με όλους αυτούς τους διαλόγους. Αλλά ίσως και πιο γρήγορα. Νομίζω πως τώρα μπορούμε να περιμένουμε λίγο γιατί μπορεί κάποιοι να έρθουν ειδικά για τις ακροάσεις. Θα κάνουμε λοιπόν πέντε λεπτάκια διάλειμμα πριν ξανακαθίσετε. Ευχαριστώ. Right, thank you everybody. Well, we have filled up a bit in the last few minutes, so I was right not to. Ε, έχουμε μαζευτεί στο μεταξύ. Χαίρομαι που δεν αρχίσαμε νωρίτερα. Θα ήθελα να καλωσορίσω το, τους τρεις α, ε, διευθυντές α, ε, των α, επαπτικών μας αρχών. Είμαστε περήφανοι για τις ευρωπαϊκές επαπτικές μας αρχές και έχουν ήδη αρκετέ εξουσίε, αν ήταν στο χέρι μα θα τι ε, ενισχύουμε ακόμη περισσότερο. Πρώτα θα μιλήσει ο Στίβεν Μάγιορ, που σε 8 λεπτά θα μας κάνει την ενημέρωση για το έργο της ε, Μικτής Επιτροπής και μετά ένα πεντάλεπτο για την ΑΚΑ και μετά ο Ανδρέα Ενρία και ο Γκαμπριέλ Μπερναρντίνο θα μιλήσουν από 5 λεπτά ο καθένας για την ε, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Πρώτα ο Στίβεν και φυσικά μετά τις παρουσιάσεις θα έχουμε και γύρω ερώτα απαντήσεων. Ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά και τα μέλη της ε, Ευρωπαϊκής ε, της Επιτροπής Κοινωνικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αποστολή της Μικτής Επιτροπής είναι να, ε, να χρησιμοποιήσει ως φόρουμ στην οποία οι υποπτικές αρχές θα ε, συνεργάζονται τακτικά και στενά για να εξασφαλίσουν διακλαδική συνοχή για πολλού τομεί. Μέσω των κοινών προσπαθειών των τριών υποπτικών αρχών του τελευταίου 18 μήνε καταλήξαμε ε, να χρησιμοποιούμε συστηματικά οι υποπτικέ αρχέ στη Μικτή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσουμε συνοχή και σύγκληση των απόψεών μα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντο, προκειμένου να καταλήξουμε σε κοινέ λύσει και να ανταλλάσσουμε πληροφορίε για του ε, διάφορου τομεί. Οι εποπτικές αρχές έχουν ε, αναλάβει τη δέσμευση και σε επίπεδο χαμηλόβαθμου και υψηλόβαθμου προσωπικού προκειμένου να επιτελέσουμε το έργο μας και να ταπεξέλθουμε στους στόχους. Ε, στόχου. Υποστηριζόμαστε στο έργο μας από τέσσερις υποεπιτροπές. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δομές αυτές. Υπάρχει Επιτροπή Κινδύνου που γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για τους κινδύνους μεταξύ των εποπτικών αρχών. Έχουμε επίσης ε, την έκθεση για, τον, για, το, για τους κινδύνους και τα τρατά σημεία του χρηματοπιστωτικού ε, συστήματος ε, μαζί με το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και φυσικά έχουμε, παρακολουθούμε, κάνουμε μια επισκόπηση της αγοράς και των προϊόντων και έχουμε και την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πρήψη, επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτε επενδυτέ. Επίση, συγκεντρώνουμε δεδομένα για τι τάσει του καταναλωτέ. Έχουμε και την υποεπιτροπή για του χρηματοπιστωτικού ομίλου, που επικουρεί την Ευρω... Ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση τη οδηγία για του χρηματοπιστωτικού ομίλου. Είχαμε φυσικά διαβουλεύσει και, με τη... και στην Μικτή Επιτροπή και η τελική μα γνωμοδότηση θα δοθεί στα τέλη του έτου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρα από τον υποεπιτροπών όμω, έχουμε και τακτικές ε, διμηνίες ε, συσκέψεις, προκειμένου να έχουμε τακτική ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις αγοράς στους διάφορους τομείς, προκειμένου να αποφύγουμε οποιαδήποτε μετάδοση των κινδύνων. Η Μικτή Επιτροπή υιοθετεί ελαστική προσέγγιση και ε, οι πρόεδροι των Αποπτικών αρχών συναντιόνται τακτικά προκειμένου να αποτρέψουν αρνητικές εξελίξεις αγοράς. Τέλος, μετά τις υποθέσεις ε, των διατραπεζικών επιτοκίων Libor και Euribor, ε, ξεκινήσαμε διάφορες εργασίες για τα επιτόκια αναφοράς και ε, μαζί με τη Μεκτή Επιτροπή ξεκινήσαμε δραστηριότητες, καταρχήν για να διευκολύνουμε τις εθνικές έρευνες ό,τι αφορά το Euribor. Δεύτερον, να προβούμε σε αναθεώρηση του συστήματος του Euribor καταλήγοντας στο σύστημα υπολογισμού των επιτοκίων και την διαδικασία υποβολής. Επίσης δίνονται κατευθυντήρες γραμμές προκειμένου να δοθούν ορόσημα συμμετοχή στην αγορά με ε, θέμα την διαφάνεια, τη σύγκρουση και τους ελέγχους και έτσι θα συμβάλλουμε στο ε, έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Και τώρα προχωρώ στο έργο και τις δραστηριότητες ε, της ε, ΕΑΚΑ ε, επικεντρώνουμε το έργο μας σε πέντε τομείς. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το ενιαίο εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το Σεπτέμβριο του 2011 είχαμε 51 ρυθμιστικά και εφαρμοστικά στάνταρ και προδιαγραφές. Ε, με αυτά τεχνικά στάνταρ έχουμε ε, για, τις, για, για τις ανοιχτές ε, πωλήσει και άλλα θέματα ρυθμιστικά τεχνικά στάνταρ. Καταρχήν θα, ε, ολοκληρώσουμε τα στάνταρ προς το τέλος του μήνα, ώστε να προβλέψουμε τους κανόνες για, τα, για τις αγορές παραγόγων μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Η ΑΚΑ έχει φροντίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμβάλλουν στην διαδικασία χάραξης πολιτικής με ανοιχτέ διαβουλεύσεις ε, επαφές ε, με ενώσεις ε, ενδιαφερομένων, παιδιτών, συμμετεχόντων στην αγορά και ζητούμε φυσικά τη γνώμη και των εμπλεκομένων στην αγορά. Και για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά το εχειρίδιο, προωθούμε την σύγκληση των εποπτικών, των εποπτικών αρχών με διάφορους και δίνουμε έσφαση και στην οδηγία MIFID. Επίσης, ε, συμμετέχουμε ενεργά στο έργο, ε, σε έργο διεθνούς επίπεδου. Για παράδειγμα, με την, ε, συμμετέχουμε στην διεθνή, στο διεθνή συντονισμό των εξωχρηματιστηριακών παραγόντων και στην εποπτεία των οίκων αξιολόγησης. Επίσης, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και αντιμετώπιση της κρίσης. Έχουμε τακτική ενημέρωση για τους κινδύνους και τα τροτά σημεία. Έχουμε ολοκληρώσει το έργο για τους κινδύνους σε σχέση με την αγορά με, για δομημένα ε, και περίπλοκα προϊόντα, την αγορά CDS και τις σκιώδεις τραπεζικές ε, δραστηριότητες στην Ευρώπη. Επίσης θα ήθελα να τονίσω κάποιες βασικές ε, δραστηριότητες της ΑΚΑ σε περίπτωση αρνητικών εξελίξεων της αγοράς. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΜΑ ε, ε, συνήρθε το ε, καλοκαίρι για να εξετάσει τις καταστάσεις αγοράς στην Ευρώπη. Έγινε ανταλλαγή πληροφοριών για βασικές εξελίξεις της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις εθνικές αρχές προκειμένου να αξιολογηθεί που χρειαζόταν συντονισμός και τι είδους σε ό,τι αφορά την προστασία του, των επενδυτών. Ενισχύσαμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για προστασία επενδυτών χάρη σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Τον Ιούλιο του 2012 δημοσιεύσαμε δύο, δύο δέσμες κατευθυντηρίων γραμμών για την ενίσχυση των, ε, των επενδυτών. Επίσης, ε, ε, δώσαμε συμβουλές για τη MIFID και το θέμα της συμμόρφωσης με τη MIFID. Τον Ιούλιο είχαμε κατευθυντήριες γραμμές για τα EDF και άλλα θέματα ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να εναρμονίσουμε τις ρυθμιστικές πρακτικές για το πολύ σημαντικό τομέα των ΟΣΕΚΑ, ε, αυξάνοντας το επίπεδο και την ποιότητα των πληροφοριών. Και μάλιστα αυτή τη βδομάδα θα ε, έχουμε κατευθυντήριες γραμμές για τις αποδοχές, προκειμένου ε, να ε, ευθυγραμμιστούν οι αποδοχές με, την υπο... με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων να δρουν διαφανώς ε, με επαγγελματικό τρόπο και υπευθυνότητα. Επίσης ασκούμε τις αρμοδιότητές μας και το Δεκέμβριο του 2011 είχαμε μια προειδοποίηση για το κινδύνους ε, στις, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και μάλιστα μετά από αύξηση των αιτιάσεων προς τις εθνικές αρχές και η ε, εποπτεία στους οίκους αξιολόγηση. Είναι η πρώτη φορά που ασκήσαμε τις εποπτικές μας ε, εξουσίες ε, στους οίκους αξιολόγηση. 17 τέτοιες, τέτοιοι και έχουν εγγραφεί και θα εξακολουθήσουμε να εξετάζουμε περαιτέρω αιτήσει. Σε ό,τι αφορά τις εποπτικές μας δραστηριότητες, η ομάδα μας κεντρικού Μητρώου έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε τρεις βασικούς φορείς. Η πρώτη έλεγχοι έγιναν το Δεκέμβριο του 2011 και τα πορίσματα δημοσιεύτηκαν το Μάρτιο. Η δεύτερη επιτόπια επιθεώρηση ολοκληρώθηκε στο τέλος του μήνα. Η έκθεση του Μαρτίου επισημαίνει διάφορες αδυναμίες και τομείς που χρήζουν βελτίωσης και θα υποβάλουμε και ε, προτάσεις μετριασμού του κινδύνου για κάθε οικοξιολόγησης. Επίσης, ε, είχαμε δεύτερο γύρο ελέγχων και εξετάζουμε τις αποδείξεις ε, και τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε προκειμένου να καταλήξουμε σε πορίσματα. Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις για τους οίκους αξιολόγησης και την υποπτία, έχουμε ε, φέτος θεσπίσει ένα κεντρικό μητρό προκειμένου να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά την, την οργάνωση της ΕΑΚ. Αφιερώσαμε ένα μεγάλο τμήμα των πόρων μα στην ανάπτυξη τη εσωτερική μας οργάνωσης. Από 45 υπαλλήλου το Σεπτέμβριο του 2011 περιμένουμε να ανέρθουμε σε 100 υπαλλήλου ε, στα τέλη του 2012. Χαίρομαι ιδιαίτερω και για την ποιότητα των προσλήψεων και για τι ικανότητε των προσλήψεων και των υποψηφίων. Επίση, σε ό,τι φορά τη χρηματοδότηση της ΕΑΚΑ θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα πρέπει να, ε, να καταλήξουμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης που θα στηρίζεται σε 100% κοινοτική χρηματοδότηση και όχι στη χρηματοδότηση που ισχύει σήμερα ή τουλάχιστον σε ένα συνδυασμό και των δύο συστημάτων. Σας ευχαριστώ. Τώρα στην EBA, ε στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής. Η κρίση του κρατικού χρέους είχε σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στον τραπεζικό τομέα της Ευρωζώνης και στην ενιαία αγορά. Ο ισχυρός δεσμός μεταξύ των τραπεζών και των κρατικών ομολόγων έγινε πιο στενός και οδήγησε σε ένα κατακαιρματισμό της ενιαίας αγοράς με βάση τα εθνικά σύνορα και με, οδήγησε σε μεγάλη αστάθεια των καταθέσεων σε πολλά κράτη-μέλη. Οι ανησυχίε των ε, επενδυτών οδήγησαν σε, μια, σε ένα πάγωμα της ε, τραπεζικής, ε, του τραπεζικού χρήματος που ήταν διαθέσιμο, ειδικά για δάνεια που είχαν μεγάλες περιόδους αποπληρω, αποπληρωμής. Και αυτό οδήγησε σε μια μαζική και άτακτη απομόχλευση από το, τα μέσα του 2011 η EBA ε, ζήτησε μια τρισδιάστατη προσέγγιση για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Πρώτον, ενίσχυση του κεφαλαίου των τραπεζών, ούτω ώστε να είναι πιο ισχυρέ για να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία και να περιορίσουν την απομόχλευση, ε, ευρωπαϊκέ παρεμβάσει για να υποστηρίξουμε την χρηματοδότηση των, από τι τράπεζε και να σπάσουμε τη σχέση με τα κρατικά ομόλογα και δράσει για να διορθώσουμε την κρίση του, του κρατικού χρέου ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, και μειώνοντας ε, τον κίνδυνο της αναδιάρθρωσης του χρέους. Ως εποπτικές αρχές εγκύψαμε αμέσως ε, και κάναμε κάποιες παρεμβάσεις. Ε, λάβαμε υπόψη τις συστάσεις που λήφθησαν υπόψη οι συστάσεις μας μάλλον στα μισά του 2011, ούτω ώστε να ενισχύσουμε τις τράπεζες ε, και έχουμε φτάσει σε ένα ποσό 190 δισεκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό πολύ κοντά στη σύσταση του του το φθινόπωρο του 2011. Τα μέτρα υποστήριξης ε, εγκρίθηκαν για τις ελληνικές και ισπανικές τράπεζες και θα αυξήσουν έτσι περαιτέρω αυτό το ποσό. Καταφέραμε αυτή την περίπλοκη διαδικασία εξασφαλίζοντα ότι οι τράπεζες δεν θα υλοποιήσουν το στόχο αυτό για τα κεφάλαια ε, τα ίδια κεφάλαια, μειώνοντα το δανεισμό στα νοικοκυριά και στι εταιρείε, ειδικά στι μικρομεσαίε. Επίση, έχουμε στενή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών τη χώρα προέλευση και χώρα υποδοχή, ούτω ώστε η κεφαλιακή ε, προσαρμογή να μην ε, επηρεαστεί από το ότι οι αρχέ μπορεί να είναι από την ίδια χώρα. Η EBA συνεχίζει τι προσπάθειε, ούτω ώστε να εξηγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών και οι τράπεζες θα πρέπει να κάνουν μια συντηρητική και συνεπή αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και να λάβουν δράσεις, ούτως ώστε να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία δανεισμού ε, στις ιδιωτικές αγορές η άνευ προηγουμένου ε, παροχή ρευστού διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από άλλες ε, Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες και η απόφαση να προχωρήσουμε προς την Τραπεζική Ένωση ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Η Τραπεζική Ένωση θα επηρεάσει τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής γιατί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεσμευτούμε ακόμα περισσότερα ούτως ώστε να έχουμε μια ενιαία δέσμη κανόνων ούτως ώστε να περάσουμε προς μια πραγματική ενιαία μεθοδολογία εποπτείας ε, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και με τον τρόπο και σε ό,τι αφορά το, τις δράσεις τις διορθωτικές. Ε, εάν δεν κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια, ε, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πόλωση ε, στην ενιαία αγορά ανάμεσα στην Ευρωζώνη, όπου θα έχουμε ενιαίους κανόνες, και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου θα έχουμε πολλαπλούς εθνικούς κανόνες. Η αρχή μας έκανε πολλές προσπάθειες για να προχωρήσει σε ρυθμιστικές ε, διορθωτικές δράσεις και στο να συντάξει αυτό το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. Ε, προτείναμε κάποια ε, σχέδια προτύπων σε διάφορους τομείς με βάση το CRD4-CRR ε, μας το ζήτησε η Κομισιόν και έχουμε ολοκληρώσει μια έκθεση για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει για τον δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένα σημαντικό θέμα και για σας. Έχουμε μια καλή μέθοδο εργασίας με ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας ε, με την ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, και με μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης και με μελέτη αντικτύπου. Αυτό θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τα σχέδια προτύπων όταν τα νομοθετικά κείμενα εγκριθούν. Είναι σημαντικό τώρα όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία να δεσμευτούν, ούτω ώστε να έχουμε αυστηρού και συνεπεί κανόνε με βάση τα διεθνή πρότυπα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί οι κανόνε θα αφορούν όλε τι τράπεζε και θα πρέπει ε, επιτέλου να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά μοντέλα και πολλέ κουλτούρε. Η αναλογικότητα θα είναι βασικό στοιχείο σε, αυτό, σε αυτή την προσπάθεια. Σε, πολλές, σε πολλούς τομείς είναι σημαντικό ότι ο πύχης για να αξιολογήσουμε την ε, ρευστότητα και την φερεγγιότητα των τραπεζών είναι ο ίδιος για όλες τι τράπεζε στην ενιαία αγορά. Η έντονη πίεση που αντιμετωπίζουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση στο τραπεζικό τομέα και στη μεταρρύθμιση των τραπεζικών κανόνων ε, μας ε, ανάγκασε να παραβλέψουμε λιγάκι στην αρχή τον τομέα της ε, προστασίας του καταναλωτή. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο ε, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Ε, ξέρω πολύ καλά επίσης ότι πρέπει να προοδεύσουμε σε αυτόν τον τομέα ε, και επειδή ακριβώς πρόσφατα είχαμε επεισόδια ε, καταχρηστικών πωλήσεων, ε, ατελού συμμόρφωσης με τους κανόνες ξεπλήματος του χρήματος και χειραγώγηση των όρων της αγοράς, εργαζόμαστε τώρα πιο εργοδός σε αυτούς τους τομείς, ούτως ώστε να υπάρξουν κάποιες σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα του, των υπόθηκων δανείων, ε, στον ε, υπεύθυνο δανεισμό και στη διαχείριση των υπερημεριών. Ε, θα ήθελα να μιλήσω τώρα για το, τους σπόρους μας, όπως και ο Στίβεν. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε. Θα ήθελα να σας πω ότι ο, οι ανθρώπινοι πόροι που έχουμε ε, και το όριο στο οποίο, το οποίο έχει καθοριστεί για μας, μας ικανοποιεί. Αλλά όμως τώρα σε αυτή τη φάση κρίσης ε, θα πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα προς την υλοποίηση του στόχου. Ε, δηλαδή να έχουμε τους ανθρώπινους πόρους στη διάθεσή μας που προβλέπονται για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι μέλη της Επιτροπής. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια δομή, να προσλάβουμε νέο προσωπικό, να φτιάξουμε εσωτερικό κανονισμό και διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά νομίζω πως καταφέραμε να προχωρήσουμε σε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο σύμφωνα με τους τομείς που μας έχει δώσει Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Το πρώτο τομέα, τον ρυθμιστικό, εμείς ε, εστιαστήκαμε στο να προετοιμάζουμε την σύγκληση των πρακτικών ε, που θα προκύψει με την οδηγία ε, για τη φερικαιότητα υπαριθμών 2. Έχουμε γύρω στις 15 κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε εκδώσει και επίσης δίνουμε στα πολιτικά θεσμικά όργανα τεχνική ανάλυση για τα βασικά ζητήματα που συζητούνται στο Omnibus 2. Οι δε σημειώσει που κάνουμε δείχνουν και τα σημειώματα δείχνουν ξεκάθαρα την ανεξαρτησία μας όσον αφορά τις επαγγελματικέ συντάξει μετά από δύο εκτεταμένες ε, δημόσιες διαβουλεύσεις απαντήσαμε στις προσκλήσεις της ε, Κομισιόν όσον αφορά και την ε, αναλογικότητα καθώς επίσης και τις ιδιαιτερότητες των συνταξιδοτικών ταμείων και προτείναμε επίσης μία ενίσχυση της διαφάνειας στα μέλη των συνταξιδοτικών ταμείων με τα ενημερωτικά έγγραφα. Κατόπιν για την εποπτεία εμείς διευκολύναμε μία συντονισμένη προσέγγιση από τα μέλη μας για την αντιμετώπιση της κρίσης με μία κοινή προσέγγιση για να παρακολουθούμε το μίσο όπως η έκθεση σε ε, τραπεζικό χρέος και χρέος ε, δημόσιο, τη ρευστότητα και τα ταμιακά διαθέσιμα, την διασύνδεση μεταξύ του ασφαλιστικού και του τραπεζικού τομέα, παραδείγματο χάρη μέσω ΣΟΑΠ και ΡΕΠΟΣ, καθώ επίση και σχέδια εκτάκτου ανάγκη. Επίση, αρχίσαμε να συντάσσουμε ένα εγχειρίδιο για τις εποπτικές αρχές για την ε, οδηγία Φερεγγιότητα 2 που συμπεριλαμβάνει τις βέλτιστες πρακτικές και θα βοηθήσει την ε, εφαρμογή ενός πιο συνεπούς πλαισίου τρίτον για την προστασία των καταναλωτών και την καινοτομία στο χρηματοοικονομικό τομέα μαζί με την έμφαση η οποία δίνεται από τον κανονισμό μας έχουμε ως στρατηγική προτεραιότητα και την προστασία των καταναλωτών και την καινοτομία και αυτό φαίνεται και από τους πόρους που έχουμε αφιερώσει σε μια σε εξειδικευμένη ομάδα στο οργανόγραμμά μα και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έχουμε κάποιε πρώτε κατευθύνσει γραμμέ, οι οποίε αναπτύχθηκαν ειδικά στον τομέα προστασία των καταναλωτών. Αυτό αφορά την αντιμετώπιση παραπώνων από, από ασφαλιστικά ταμεία και ε, θα έλεγα πως καλύπτει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρυθμιστικό κενό και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά την πώληση ασφαλιστικών συμβολέων. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής μας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, το Δεκέμβριο θα οργανώσουμε την δεύτερη ημερίδα μας για την στρατηγική των καταναλωτών και θα εξηγήσουμε την ε, σχετική μας στρατηγική και τις προτεραιότητες μας τέταρτον για την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Βεβαίω, εργαζόμαστε εδώ πέρα σε τριμηνιαία βάση, αξιολογούμε την θέση μας με ποιοτικού και ποσοτικούς δείκτες για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την εξέλιξη των κινδύνων στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Επίσης υπάρχει ένα εναρμονισμένο πανευρωπαϊκό stress test το οποίο δείχνει πως ο κλάδος θα επηρεαστεί αρνητικά εάν υλοποιηθεί ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο αποδόσεις θα παρέμειναν χαμηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα κατόπιν στον τομέα των διεθνών σχέσεων πέραν των ε, επαφών και αξιολογήσεων που έχουμε σε τρίτες χώρες με βάση την οδηγία για τη φεργιότητα 2 έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τρίτες χώρες αναλύοντας και το τι γίνεται στα καθεστώτα Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα Βεβαίως, κορυφαίο ρόλο σε αυτό παίζουν οι δύο ομάδες μας οι οποίες είναι η ομάδα ασφαλιστών και αντασφαλιστών και βεβαίως η ομάδα ενδιαφερομένων ασφαλισμένων που αποτελούν βασικό μέρος της δουλειάς μας. Όσον αφορά τον προπολογισμό και τους πόρους, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στήριξη σε αυτή την ε, διαδικασία για τον προπολογισμό του 2013 και βεβαίως μέσα στα πλαίσια που επιβάλλει η τωρινή κρίση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε ένα επίπεδο χρηματοδότηση ανάλογα με τη φιλοδοξία του έργου αυτού και θεωρώ πως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία οποιαδήποτε νέα καθήκοντα μας ανατεθούν να συνοδευτούν και από τους ανάλογους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ανεξάρτητη λειτουργία μας και θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάτι το οποίο θεωρώ πως είναι σημαντικό. Αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσληψη εμπειρού προσωπικού. Αυτό το αναγνώρισε παραδείγματο χάρη και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Κομισιόν. Κατά την άποψή μας αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να έχουμε μια πιο ευέλικτη εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο συνολικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Όπως είπα, πέρσι εγώ θα προτιμούσα μια χρηματοδότηση από μια ξεχωριστή γραμμή στον προπολογισμό τη Ένωση για να διασφαλίσει την εξαρτησία μα. Τέλο, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, θέλω να τονίσω το ότι πρέπει να μπουν στην οδηγία ασφαλίσεων και συντάξεων διατάξεις που θα περιορίζουν τι ε, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, αλλιώς το άρθρο 9 δεν έχει πάρα πολύ νόημα. Κατόπιν οι επαγγελματικέ συντάξει, ο λεγόμενο δεύτερο πυλώνα, θεωρώ πως ε, αν είναι να εφαρμοστεί σωστά η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για επαρκή συντάξει, σημαίνει πω θα πρέπει να υπάρχει και ε, μια επαρκή στήριξη του λεγόμενου τρίτου πυλώνα, των ε, ιδιωτικών ε, συντάξεων, στον οποίο θα πρέπει να επεκταθεί και η αρμοδιότητά μας, κάτι το οποίο προτείνει και η αρμόδια ομάδα Είμαι σίγουρος πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να μας υποστηρίζει. Κάνουμε πραγματικά πολύ καλή δουλειά για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να χωρέσουν όλα αυτά σε λίγα λεπτά. Είμαι σίγουρος πως θα κάνουν οι βουλευτές κάποιες ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν. Εάν όχι μπορείτε να μας το πείτε. Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα τους ε, συντονιστές και μετά και τη Πέρα λοιπόν από τους συντονιστές έχω στον κατάλογο την άλλη ποδηματά, Πίτερ Σκίνερ, τον Ήβα στη Δίκη Φόρντ και τον κύριο Λουτβίξον. Άντελιν. Okay, right, that's fine. Ωραία. Ζαμπόλ, λοιπόν. Merci, Madame la Ευχαριστώ. Σας προειδοποιώ ότι δεν πρόκειται να θέσω ερωτήσεις. Θα ήθελα απλώς να πω στους τρεις ε, πρόεδρους ε, ότι εκτιμούμε ιδιαίτερο στο έργο τους και έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εξαιτία των πενιχρών ε, ε, δημοσιονομικών ε, υλικών και ανθρώπινων πόρων για να ανταπεξέλθουν στο έργο τους. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τις ευρωπαϊκές ε, εποπτικές αρχές, θυμάμαι ότι τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ταχθεί πέραν εξάρτητων εποπτικών αρχών το είπε ο κύριος Μπερναντίνο, ότι θα πρέπει να έχουν τα μέσα, τους πόρους και τις αρμοδιότητες. Βέβαια, ελάχιστε ήταν οι που έκαναν ε, τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό και σήμερα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την Τραπεζική Ένωση, μια πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, που έγινε πριν από δύο χρόνια. Βέβαια, είπαμε τις προάλλες ε, στην Ολομέλεια στον Επίτροπο Μπαρνιέ ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκινάνε είναι πολύ επικίνδυνες, γιατί αν μετά τις αναγγελίες ε, που έγιναν δεν καταλήξουμε ε, σε υπέρβαση των κοντόφθαλμων εθνικών συμφερόντων χάρη ενός συλλογικού ευρωπαϊκού συμφέροντος, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και αυτό θα είναι πολύ σοβαρό και απογοητευτικό. Πάντως το ΕΛΚ, ε, όπως φάνηκε στην ψηφοφορία για του, τον προπολογισμό θα υποστηρίξουμε ενίσχυση των πόρων ε, των ε, εποπτικών αρχών. Μερικές φορές ε, ήμασταν κάπως αυστηροί απέναντι σε κάποιες εποπτικές αρχές. Φυσικά περιορίζεστε από την εντολή σας και από τις εξουσίες και αρμοδιότητές σας. Και στο μέτρο που δεν έχουν ενισχυθεί εξουσίες σας δεν μπορείτε να αναλάβετε και περαιτέρω αρμοδιότητες. Πάντως έχουμε εδώ ένα κοινό αγώνα, μια κοινή μάχη, γιατί είναι προς το κοινό μας συμφέρον οι εποπτικές αρχές να διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο τους και να έχουν και τα, τις ικανότητες και τα μέσα, ώστε να μην μετατραπούν σε αποδιοπομπαίο τράγο όταν συμβεί κάτι να λέει «Α, η εποπτική αρχή δεν ανταπεξήλθε στο έργο της», ενώ ούτε νομικές αρμοδιότητες είχε για κάτι τέτοιο, ούτε πόρους και απλώς... α η εποπτικη αρχη δεν ανταπεξηλθε στο εργο της ενω ουτε νομικες αρμοδιοτητες ειχε για κατι τετοιο ουτε πορους και απλως ήταν το εξηλαστήριο θύμα. Αυτά και συνεχίστε στο δρόμο που χαράξετε. Ε, εμείς θα σας προσφέρουμε την αμέριστη υποστήριξή μας και την βοήθειά μας. Όπως είπες, δεν έκανες καμία ερώτηση, οπότε ας προχωρήσουμε στην Ελίζα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους ε, τους Προέδρους, ε, με κάλυψε πολλά σημεία ο συνάδελφος Γκοζές. Εγώ θα επικεντρωθώ σε τρεις ερωτήσεις. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες για εναρμόνιση των κανονισμών και των τεχνικών ρυθμιστικών προδιαγραφών. Αυτό λειτουργεί τώρα σε... στη φάση της εφαρμογής. Δηλαδή, εφαρμόζονται και εμπράκτος αυτές οι ρυθμίσεις και οι κανόνες προκειμένου να μην ε, τεθεί να αφιβόλω η λειτουργία της ε, ενιαίας αγοράς. Η ΕΙΟΠΑ θα αποτελέσει ε, με βάση το άρθρο 127.6 θα αποπτεύσει τις τράπεζες μόνο και όχι τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τι γίνεται όμως ε, με μια τράπεζα που έχει και ασφαλιστικές εταιρείες αφού είστε αρμόδιοι μόνο για την εποπτεία των τραπεζών. Δεύτερη ερώτηση. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις της προσαρμογής της ΕΤΑ στο, στη νέα πρόταση για την Τραπεζική Ένωση για να αποφευθούν αντιφάσεις και συγκρούσεις. Η, τα stress test, οι προσωμιώσεις ακραίων συνθηκών μας έδωσαν μια πρώτη εντύπωση και ήταν μια προκαταρκτική εργασία. Ποια ήταν όμως τα τροτά σημεία αυτής της προσπάθειας και τι μπορεί να βελτιωθεί για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες αν απαντούμε μεμονωμένα τις ερωτήσεις. Καλύτερα να συγκεντρώσουμε μερικές ερωτήσεις για να απαντηθούν μαζικά, συλλογικά. Ποιος θέλει το λόγο από τους φιλελεύθερους, Σιλβί. Σύντομα, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους ομιλητές για όλους όσους, όλα όσα μας είπαν και όσα κάνουν. Ε, θέλω να αναφερθώ και σε αυτά που είπε η Ελίζα λιγάκι. Αυτές τις νέες προτάσεις, τι άποψη έχετε για αυτές. Παραδείγματο χάρη συνδυασμό τραπεζών και ασφαλίσεων, ασφαλιστικών οργανισμών. Πώς συνδυάζεται το έργο της ΕΙΟΠΑ με το έργο της ΕΤΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ηρεμήσει λίγο η συζήτηση και να δούμε έτσι με ηρεμία τι άλλαξε. Τελικά θέλουμε περισσότερη ευρωπαϊκή εποπτεία. Δεν είμαστε κατά. Ο κύριος Ανδρέας ε, θα μας πει ε, πώς ε, συνδυάζεται το έργο της ΕΟΠΑ και της ΕΤΑ. Θέλω να απαντήσετε τους ώστε να καθησυχάσετε και τους συναδέλφους από χώρες που δεν είναι της Ευρωζώνης. Σε αυτή τη φάση χρειαζόμαστε την τεχνογνωσία σας. Να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα, γιατί είναι εύκολο να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου. Αλλά, κύριε Ενδρία, τι θα γίνει για τις τράπεζες ε, οι οποίες βρίσκονται κάπου μεταξύ ε, της Ευρωζώνης και των χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Ακόμα ένας και μετά θα απαντήσουμε. Η ΚΕΙ. Οκ, η ΚΕΙ. Ευχαριστώ. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση προς την Έσμα Καλωσορίζω λοιπόν τις κατευθύνες γραμμές σας προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές για ζητήματα που φορούν τι αγορές το τελευταίου έτος και πολλές από αυτές είναι πάρα πολύ λεπτομερείς και βοηθάνε πάρα πολύ και πραγματικά έγιναν δεκτές με ευχαρίστηση από τις αρμόδιες αρχές. Τώρα όσον αφορά τις συζητήσεις του δεύτερου επίπεδου που γίνονται αυτή τη στιγμή ε, σε ζητήματα όπως ο Εμίρ, είστε πάρα πολύ κοντά στην προθεσμία. Ποια διαδικασία υπάρχει ως καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη και έχει δικαίωμα να εξετάσει τι ε, τεχνικές σας ε, προτάσεις. Ποια, με ποια διαδικασία φαντάζεστε ότι θα εμπλακούμε, πώς ακριβώς θα εκπληρώσουμε τον ε, ρόλο μας ως συνομοθέτης και όχι ως ένας απλός ενδιαφερόμενος. Κάποιοι το καλοκαίρι μας περιέγραψαν ως ένα ενδιαφερόμενο μέρος. Ελπίζω και θεωρώ ότι είμαστε κάτι παραπάνω και μια κάπως... Ε, αυτά δύο ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Πόσο σίγουροι είστε πως οι τεχνικές προδιαγραφές ε, τις οποίες ε, βγάζετε στο τέλος του μήνα θα γίνουν κτές από εμάς και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Καλύτερο είναι νομίζω να μείνουμε στη σειρά που είχαμε, ξεκινώντας με την ΕΣΜΑ. Ο Αντρέα μετά έχει αρκετά να απαντήσει και μετά ο Γκαμπριέλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Φερέιρα για τις ερωτήσεις του. Για το πώς λειτουργούν τώρα τα τεχνικά πρότυπα και πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Βλέπετε στα, στις εργασίες του περασμένου έτους ότι δώσαμε έμφαση στο ενιαίο εγχειρίδιο. Λογική συνέπεια της ε, ρυθμιστικής μεταρρύθμισης ε, που είναι να εξελίξει. Κάποια στιγμή λοιπόν είναι σημαντικό όμως να έχουμε και επαρκείς πόρους και για τα άλλα κομμάτια της δουλειάς μας. Τώρα ασχολούμαστε κυρίως με το ενιαίο εγχειρίδιο, το ξέρουμε. Όμως η ΕΣΜΑ δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με το εγχειρίδιο, αλλά και με την εποπτεία και την άμεση εποπτεία. Και η εποπτεία των οίκων αξιολόγησης είναι μια δουλειά που πάει καλά. Αλλά η συμμόρφωση και η συνέπεια ε, θα πρέπει να είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει όταν προχωρήσουν και τα τεχνικά πρότυπα. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε τη 12 περίοδο για τα τεχνικά πρότυπα. Ε, για το ΕΜΙΡ είχαμε 7 μήνες για το short selling είχαμε 4-5 μήνες. Είναι δύσκολο για την ΕΣΜΑ, αλλά είναι δύσκολο και να εξασφαλίσουμε την εμπλοκή της αγοράς. Γιατί μόνο έτσι θα γίνουν αποδεκτά τα πρότυπα, αν εμπλακεί και η αγορά. Νομίζω ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση. Με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές προτάσεις είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε το δεκάμινη περίοδο ολοκλήρωσης των τεχνικών προτύπων για το ΕΜΙΡ. ήταν το πιο σημαντικό θέμα που μας απασχόλησε το 12. Τεράστια δουλειά απαιτούσε. Και την κάναμε. Έχουμε μια καλή ομάδα που ασχολείται με το ΕΜΙΡ. Είμαι, ε, έχω εμπιστοσύνη έτσι, στην δουλειά που κάνουμε. Είναι ποιοτική και σίγουρα μας πίεσε πάρα πολύ. Η ομάδα αυτή ασχολήθηκε νυχθημερών με το θέμα του ΕΜΙΡ. Δεν είναι εύκολο να περιμένουμε, να προβλέψουμε την τελική απόφαση. Λαμβάνεται μερική πλειοψηφία, αλλά ούτως ή άλλως πιστεύω ότι θα είμαστε εμπρόθεσμοι. Ξέρω ότι είστε εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία ολοκλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών. Έχετε το δικαίωμα να παρέμβετε ούτως ή άλλως, να πείτε τις απόψεις σας και εμείς εν συνεχεία θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές. Επίσης μην ξεχνάμε και ότι θα πρέπει να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις του G20. Να είμαστε έτοιμοι την άνοιξη δηλαδή, του 2013. Για την Τραπεζική Ένωση, οι περισσότερες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τους δύο συναδέλφους. Το μόνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι συνεργάζονται οι εποπτικές αρχές για τα αξιόγραφα και τις αρχές σε εθνικό επίπεδο. Πολλές ε, τράπεζες συμμετέχουν στην αγορά, έχουν εταιρείε με περιουσιακά στοιχεία, συμμετέχουν στις υποδομές της αγοράς, υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις εποπτικές αρχές των αξιογράφων και την ε, προνοιακή εποπτεία. Φυσικά αυτά πρέπει να οργανωθούν σωστά Είναι πολύ σωστό που στην πρόταση υπάρχει η προϋπόθεση να συνεργαστούμε οι τρεις αρχές και η ΕΣΜΑ. Αλλά θα πρέπει αυτή η συνεργασία να πάρει πραγματικά σάρκα και οστά. Ο Ανδρέα. Ευχαριστώ. Πρώτο σημείο για την προσπάθεια εναρμόνισης των κανόνων. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για την εναρμόνιση των κανόνων. και εσείς και εμείς με το CRD4, CRR. Αλλά είμαστε κάπου στα μισά του δρόμου. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα δεδομένα των τραπεζών στην προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Θα πρέπει να φτιάξουμε έτσι ένα μέσο όρο, μια μέση ας πούμε ευρωπαϊκή τράπεζα και μετά εφαρμόζουμε την πιο περιοριστική και την πιο χαλαρή ε, προσέγγιση σε τρεις-τέσσερις ε, τομείς όπου υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και η διαφορά είναι 300 ε, μονάδες βάσης. Πολλά πρέπει να κάνουμε ακόμα για να εναρμονίσουμε τους κανόνες λοιπόν. Τούτου λεχθέντος, ακόμα και όταν έχουμε τους ίδιους κανόνες, σε εθνικό επίπεδο έχετε πολύ διαφορετικές μεθοδολογίες για αξιολόγηση των ε, κινδύνων της τράπεζας και για να ε, δρομολογήσει στην διορθωτική δράση. Δηλαδή με τους ίδιους κανόνες μπορεί να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα. Κάναμε αυτά τα τεστ αντοχής, την προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο πακέτο για την Τραπεζική Ένωση. Ένα ενιαίο εγχειρίδιο για τους εποπτικούς κανόνες. Στις ΕΠΑ, ε, τέλος της δεκαετίας ε, έδωσα την εντολή σε όλες τις αρχές να ετοιμάσουν ένα εγχειρίδιο το οποίο θα είχαν μαζί τους αναχείρας όταν κάνανε επισκόπηση των τραπεζών. Και το ίδιο πρέπει να κάνουμε εμείς στην ενιαία αγορά. Όχι μόνο στην Ευρωζώνη, αλλά στην ενιαία αγορά. Τα τεστ αντοχής, οι δοκιμές αντοχής. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ακούστηκαν πολλές επικρίσεις για αυτά τα τεστ. Νομίζω ότι κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια όμως για να εξασφαλίσουμε τη συνέπεια στα δεδομένα που λαμβάνουμε, να πιέσουμε για αύξηση του κεφαλαίου τη στιγμή που πραγματικά το χρειαζόμαστε. Ε, το κεφάλαιο που εγχύθηκε, που ρίχτηκε στο σύστημα, ήταν τρει φορές υψηλότερο από το κεφάλαιο που έπεσε το 2009 στις ΗΠΑ. Η ενίσχυση δηλαδή του συστήματος ήταν απίστευτη. Όμω, είχαμε και κάποιες αρνητικέ συνέπειες, γιατί σε ορισμένε περιπτώσει είχαμε τράπεζε που πέρασαν το τεστ, είχαν ελάχιστα προβλήματα στο τεστ και μετά από λίγες εβδομάδες ή μήνες ας πούμε χρειάστηκε να συγκεντρώσουν περισσότερο και άλλο κεφάλαιο. Ε, το χάρη Ντέξια και η Μπάνκια. Αν λοιπόν ε, δίνουμε την ευθύνη για τα τέστ test, θα πρέπει να υπάρχει και νομική ευθύνη ότι τα αποτελέσματα είναι αξιόπιστα. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση, δηλαδή, να πηγαίνουμε στι τράπεζες, να ερχόμαστε σε επαφή άμεση μαζί του και να είμαστε σίγουροι ότι τα δεδομένα που μας δίνουν είναι αξιόπιστα. Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή, δυστυχώ. Τραπεζική Ένωση, τελικό σημείο. Θέλω να σα πω καταρχά ότι το τελευταίο που θέλω είναι να μπούμε σε μια διελκυστίδα μεταξύ τραπεζών. Πρέπει να γίνει τώρα η Ένωση και γρήγορα. Γιατί η διασύνδεση μεταξύ των τραπεζών και των κρατικών ομολογών, δημιουργεί κατακαιρματισμό στην αγορά. Δημιουργεί τεράστιους κινδύνους. και δημιουργεί ε, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πρέπει να γίνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και μάλιστα με φιλόδοξο τρόπο. Φυσικά. Υπάρχουν προκλήσεις και στη σχέση μεταξύ της ΕΚΤ και της ΕΤΑ. Δεν είναι εύκολη λύση. Οι προκλήσεις αυτές αφορούν το πώς θα βρούμε την κατάλληλη κόλλα για να μείνει ενιαία η αγορά. Θα πρέπει η ΕΚΤ να κινηθεί γρήγορα σε ενιαίους κανόνες. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε τις τράπεζες ας πούμε, με διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με το, τη χώρα από την οποία προέρχονται, που βρίσκονται εγκαταστημένες και η νομοθεσία που είναι ενώπιόν σας δυστυχώς αφήνει μεγάλο περιθώριο εθνικής ευελιξίας. Μπορεί να έχουμε δηλαδή ενιαίους κανόνες στην Ευρωζώνη και ευελιξία για την υπόλοιπη ενιαία αγορά. Και αυτό θα οδηγήσει σε μια πόλωση φυσικά. Το δεύτερο σημείο είναι οι εποπτικές πρακτικές. Η ΕΚΤ θα πρέπει να πιέσει ούτως ώστε η εποπτεία να ασκείται με ενιαίο τρόπο στην Ευρωζώνη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να γίνει αυτό και σε επίπεδο ενιαίας αγοράς. Δηλαδή να κινηθούν προς την, κατή, προς την ίδια κατεύθυνση, ίδια μεθοδολογία. Ε, πραγματικά συνεπή προσέγγιση. Συνολικά η ενιαία αγορά, όχι μόνο η Ευρωζώνη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά θέματα. Και στο μέλλον μην ξεχνάμε Και το θέμα της εξυγίασης. Βασικό θέμα. Ε, οι επενδυτές κοιτάνε τις τράπεζες α, και ψάχνουν να βρουν τα κρατικά ομόλογα που θα τους δώσουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Όσο πιο ολοκληρωμένη ενιαία είναι η εσωτερική αγορά, τόσο περισσότερο ανθεκτική θα είναι η Ένωση. Αυτά είναι τα βασικά ε, θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, καθώς ε, δημιουργούμε, χτίζουμε την Τραπεζική Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να αναφερθώ και εγώ σε αυτά τα δύο στοιχεία. Βεβαίω, στον ασφαλιστικό τομέα, το ζήτημα των προτύπων και των κανόνων και των εποπτικών πρακτικών έχει τεράστια σημασία και εγώ λέω πως εάν πιστεύουμε πως με το να έχουμε ενιαίους κανόνες θα έχουμε λύσει όλα, κάνουμε λάθος. Πρέπει να υπάρχουν πιο ενιαίες πρακτικές επίβλεψης, εάν είναι να έχουμε εσωτερική αγορά. Και βεβαίω ε, στην ασφαλιστική αγορά εργαζόμαστε σκληρά για την οδηγία για τη φρικιότητα 2 και ελπίζουμε να την έχουμε συντομότερα γιατί έτσι θα έχουμε ενιαίους κανόνες. Έχουμε πράγματι όπως είπα όλες αυτές τις προδιαγραφές και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν μεγάλη σημασία αλλά ακριβώ επειδή θεωρούμε πως η εποπτεία και η όμοια υποπτία, η ομοιόμορφη υποπτία είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Αν δείτε παραδείγματο χάρη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτική σταθερότητα αμέσω μετά την κρίση βεβαίω μιλάνε για υψηλό βαθμό φερεγκαιότητα κεφαλαίου, μιλάνε για τη λύση τραπεζών, μιλάνε για καλύτερη διαχείριση του κινδύνου, αλλά μιλάνε και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξεχνιέται λίγο. Οπότε αυτό έχει κέρια σημασία και θα πρέπει νομίζω και σε διεθνές επίπεδο να κάνουμε μαθήματα ως προς αυτό. Γι' αυτό και η εφαρμογή έχει ουσιαστική σημασία. Γι' αυτό στην ΕΙΟΠΑ αρχίσαμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα για να αναπτύξουμε αυτό το, να αναπτύξουμε αυτό το εγχειρίδιο, όπως το λέμε, που ξεκινάει με τις βέλτιστες πρακτικές στον κάθε τομέα και μετά βήμα-βήμα θα καταλήξει να είναι το εγχειρίδιο, όπως είπα, για αυτούς τους ε, στόχους, στόχους υποκτίας. Πρέπει να γίνει αυτό για την ενιαία αγορά. Δεύτερον, για την Τραπεζική Ένωση. Εγώ, ως ε, άνθρωπος ο οποίος πραγματικά πιστεύει στην Ευρώπη, θεωρώ πως κάνουμε όντως ε, τι σωστέ πράξει. Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο υποπτικός μηχανισμό στην Ευρώπη, αλλά βέβαια οι ασφάλειες δεν είναι τράπεζε. Έχουμε διαφορέ διαφορές ε, κινδύνους, διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη ε, συνέπεια. Τώρα, εγώ δεν θέλω να μπω στο θεσμικό ζήτημα, αν πρέπει να είναι η ΕΚΤ ή η ΕΟΠΑ κτλ. Το βασικό για εμάς είναι να γνωρίσουμε πως και στον τομέα των ασφαλιών πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η διαδικασία για, για να το σκεφτούμε λίγο, να το αναλογιστούμε κι εμείς, να δούμε δηλαδή ποια βήματα θα πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τα καθήκοντα της αρμοδιότητας σε ΙΟΠΑ στον τομέα της εποπτείας και σας βεβαιώ πως θα καταθέσουμε κάποιες ιδέες, τις εξετάζουμε, υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε και θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιομορφία. Βεβαίως ε, πρέπει να υπάρχει και υποπτία των διασυνοριακών ομίλων. Μετά για το ερώτημα των ε, χρηματοπιστωτικών ομίλων. Πράγματι πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι για το τι περιέχει εδώ πέρα η Κομισιόν για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Και πως υπάρχει αυτός ο περιορισμός από τη συνθήκη για την εποπτεία ασφαλιστικών εταιριών, αλλά υπάρχει η πραγματικότητα των χρηματοπιστωτικών ομίλων, οπότε πρέπει να είναι τα πράγματα πιο ξεκάθαρα και βεβαίω υπάρχουν προκλήσεις για το πώ θα εφαρμοστεί η Τραπεζική Ένωση στου χρηματοπιστωτικού ομίλους. Πρέπει να υπάρξει εκεί πέρα νομίζω ένα ρόλος για να υπάρχει ακριβώς ενιαία εποπτεία εντό τραπεζική Ένωση, αλλά ε, ελπίζουμε να ε, εξεταστεί όπως σας είπα και ο τομέας των ασφαλείων. Λοιπόν, θα ακούσουμε του επόμενου τρει: Σβέν, Γιούργεν και την Άννη Ποδηματά. Σβάν. Μπορεί να μην σας βλέπω γιατί έχει μπροστά σας ο κάμεραμαν και κάμερα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε και θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια. Ευχαριστώ και για τις γραπτές απαντήσεις που μας στείλατε. Βέβαια, εξακολουθώ να έχω πρόβλημα με τη σύνθεση κάποιων ομάδων ενδιαφερομένων. Δεν μου δόθηκε και σαφής απάντηση γι' αυτό. Επίσης, είχα κάποιες κακές εμπειρίες τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα, αναλογική εκπροσώπηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης ε, και υποβολή εκθέσεων σε τράπεζες ε, και τον τρόπο που κρατάν ε, τα λογιστικά του στοιχεία. Και μια και έχουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση, φαντάζομαι ότι για όλους τους ενδιαφερόμενους εξευρωπαϊσμός δεν σημαίνει ότι εξαλείφεται η ποικιλομορφία είμαστε υπέρ της φιλοευρωπαϊκής γραμμής που ταυτόχρονα όμως θα λαμβάνει υπόψη και την διαφορετικότητα και θεωρεί ως πλούτο την ποικιλομορφία και δεν θα συγχαίουμε την ποικιλομορφία με την ελαστικότητα, την υπερβολική επίοικια ή την ελαστικότητα ως προς τις αδυναμίες. Σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση. Ε, δεν ήταν αρκετά ισχυρά αυτά που ακούσαμε και αυστηρά για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Θα έπρεπε να ήσασταν πιο κατηγορηματικό, κύριε Μπερναντίνο. Ποιο είναι ο ρόλο τη ΕΙΟΠΑ και τι ακριβώ θέλετε, τι δικαιώματα, τι κανόνε, τι δομέ. Και τέλο. Θέλω να μας πείτε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες τι προβλήματα αντιμετωπίσατε στο έργο στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο έργο των εθνικών εποπτικών αρχών. Γιατί δεν θα πρέπει να κολλήσουμε στα ίδια προβλήματα και στην τραπεζική έντονση με αυτά που αντιμετωπίσαμε στα stress test. Είπατε, θέλετε πρόσβαση, άμεση πρόσβαση στα δεδομένα, κυρία Ερία, και δυνατότητα πραγματοποίηση ελέγχων. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Αντιμετωπίσατε προβλήματα και στις άλλες εποπτικές αρχές, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Και τι δομές χρειαζόμαστε για να υπερκεράσουμε τέτοια προβλήματα και έχω μεγάλη περιέργεια. Τι δραστηριότητε θέλει να αναλάβει η ΕΤΑ σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Γιατί από τα τρία θεσμικά όργανα εσείς το αναφέρατε και μέχρι στιγμής ήταν οι πιο, χαρα... πιο... που περισσότερο στο θέμα αυτό και ελπίζω να μου πείτε ποια θα είναι τα επιπλέον βήματα. ναι, πολλά ήδη ακούστηκαν θα ήθελα και εγώ να πω ορισμά. Η συνεργασία, έχετε δύο επίπεδα συνεργασίας, ένα οριζόντιο μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και η κάθετη ε, συνεργασία μεταξύ ημών δηλαδή και των εθνικών αρχών. Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω πού βλέπετε κενά, πού θα λέγατε πως κάπου πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει συγκεκριμένα. Δεύτερον, το δεύτερο ερώτημα το οποίο το απευθύνω και στους τρεις σας. Τα μέσα τα οποία σας έδωσε η πολιτική για να κάνετε τη δουλειά σας επαρκούν είναι αρκετά ή θεωρείτε πως θα πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Είμαστε σε μια φάση όπου δοκιμάζουμε πως λειτουργούν τα πράγματα. Ακόμα ξεκινάμε, οικοδομούμε. Οπότε το ερώτημά μου είναι αυτό. Τι θα θέλατε εσείς να βελτιωθεί. Τώρα, για την Τραπεζική Ένωση, ο Ανδρέα είπε ήδη κάποια πράγματα, αλλά εγώ παρόλα αυτά θα ήθελα να ρωτήσω. Έχει νόημα να, υπάρχει, να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός της ε, εποπτείας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της ε, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής έχει νόημα σε μια ενιαία αγορά να το σπάσουμε σε δύο επίπεδα. Και τελευταία συγκεκριμένη ερώτηση προς τον κύριο Μπερναρντίνο σε γερμανικά μήμια διάβασα πως θα καθυστερήσει ακόμη μία φορά η εφαρμογή της οδηγίας για τη φερικιότητα 2. Θα ήθελα να μάθω πώς το βλέπετε εσείς. Um, I think it's Annie. Yes. ναι. Thank you, Sharon. Thank you, chairs. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους Πρόεδρους των υποπτικών Αρχών Ε, μία αποτελεσματική εποπτική, ε, τραπεζική υποπτία θα αποτρέψει όχι μόνο μελλοντικέ κρίσει, αλλά θα εξασφαλίσει και κατάλληλη χρηματοδότηση τη πραγματική οικονομία. Έχω μία ερώτηση προ τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Καταρχήν, βέβαια, θα πολύ ευχαρίστω να ακούσω τα σχόλια και των άλλων δύο πρόεδρων. Κύριε Ενρία, επανέρχομαι στην σύσταση των τελών του 2011 που απαιτούσε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών Εκεί επισημέναμε ότι οι κεφαλικές ελλείψεις των τραπεζών εμπόδιζαν την δυνατότητά τους να συγκεντρώσουν χρήματα, κάτι που δημιουργούσε ύφεση ε, στην πραγματική οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση τα στοιχεία σα 95% των προβλημάτων που εντοπίστηκαν, αντιμετωπίστηκαν από τις ε, δράσεις άμεση χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά η πρόσβαση των οικοκυριών στο δανεισμό ήταν πολύ περιορισμένη για των επιχειρήσεων. Και αναφέρθηκαν φοροαποφυγέ, ε, κάποιες κρατικέ ε, εγγυήσει, αλλά βέβαια δεν είναι και πολύ βιώσιμη αυτή η λύση εξαιτία τη φορολογική, δημοσιονομική εξηγήση. Τι πολιτικέ λοιπόν και τι εργαλεία χρειαζόμαστε ώστε να εξασφαλίσει και πάλι ρευστότητα στην πραγματική οικονομία ο τραπεζικός κλάδος και μια και θεωρείται ότι η μετάβαση προς ε, την κεφαλαία αγορά είναι, λύση. Τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα, ε, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα πρόσβαση στην κεφαλαία αγορά από ότι οι μεγαλύτερες εταιρείε. Ωραία. Θα ακούσουμε ή με την ίδια σειρά τους Πρόεδρους ή με αντίστροφη όπως προτιμάτε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε μερικά από τα σχόλια. Καταρχήν, ως προς τη σύνθεση των ομάδων ενδιαφερομένων. Στην ΕΑΚΑ εφαρμόσαμε μια πολύ αυστηρή διαδικασία για να καταλήξουμε στην πιο σωστή σύνθεση. Είχαμε βέβαια περιορισμένη διακριτική ευχέρεια σε ό,τι αφορά την γεωγραφική εξορόπηση που έπρεπε να λάβουμε υπόψη για την αντιπροσωπευτικότητα των διαφόρων ομάδων. Οι περισσότερε αλυσίδε εκφράστηκαν για τη χαμηλή εκπροσώπηση των καταναλωτών. Πάντω, μα ικανοποίησε εμάς ε, ε, η εκπροσώπηση αυτή, γιατί στη δική μας ομάδα έχουμε πρόεδρο από την ομάδα των επενδυτών. Οπότε αν θέλουμε μεγαλύτερη ανάμεξη, γιατί ο χρηματοπιστωτικός κλάδος σίγουρα είναι ισχυρότερο και έχει και τους περισσότερους πόρους, αλλά θα πρέπει να δούμε και τη σύνθεση προβλέπει ο κανονισμός για την ομάδα των ενδιαφερομένων. Ίσως εκεί θα πρέπει να εμβαθύνετε, αν θέλετε να τροποποιηθεί η σύνθεση. Πάντως, δεδομένου του πλαισίου που μας δεσμεύει, νομίζω ότι εξασφαλίστηκε καλή εκπροσώπηση και των καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά την οριζόντια συνεργασία μεταξύ των τριών εποπτικών αρχών, νομίζω ήταν πολύ εντυπωσιακή πρόοδος ε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Βέβαια διαπιστώσαμε ότι η Μικτή Επιτροπή, ούτε είναι ούτε είναι πρόθεσή μα να γίνει το πρόσωπό μας προς τον έξω κόσμο. Από αυτή την άποψη έχουμε μπει σε μια κανονική πορεία σε ό,τι αφορά την οριζόντια συνεργασία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, αλλά κατά τη γνώμη μας το επίπεδο στο οποίο καταλήξαμε και που φτάσαμε είναι ικανοποιητικό. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ της ΕΑΚΑ ε, και τη συνεργασία των υπαλλήλων της ΕΑΚΑ με τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές, Τώρα, προτείναμε να περάσουμε σε πλήρη κοινωτική χρηματοδότηση ή σε μηχανισμό που θα προέρχεται από τη βιομηχανία. Ε, ενώ τώρα έχουμε συγχρηματοδότηση και από τα κράτη-μέλη. Ε, όταν ψήφισαν τα κράτη-μέλη περισσότερε αρμοδιότητε για την ΕΣΜΑ, ουσιαστικά πλήρωσαν, ε, ψήφισαν και χαμηλότερο προπολογισμό για, τους, για τα ίδια τα κράτη-μέλη. Και το επαπτικό μα σύστημα δεν είναι σύστημα που θα παίρνουμε από το εθνικό επίπεδο και θα ενισχύουμε το ευρωπαϊκό, αλλά που θα ενισχύουμε και τα δύο επίπεδα. Οπότε από αυτή την άποψη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται σε πολύ δύσκολη ε, θέση όταν πρέπει να ψηφίζουν ε, ενισχυμένο προπολογισμό ε, για την ΕΣΜΑ, ενώ σε εθνικό επίπεδο έχουν προβλήματα οικονομικά, έχουν τον ΕΜΙΡ, τη ΜΥΦΙΤ και εκεί αυξάνονται επίσης οι ευθύνες τους και το έργο τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κλαδική, την κλαδική τομεακή νομοθεσία, Θέλουμε φυσικά να ενισχυθεί η προστασία του καταναλωτή και μπορούμε να ενισχύσουμε την εποπτεία μας, αλλά θα πρέπει και η τομεακή νομοθεσία να μας βοηθά. Βέβαια η δεύτερη οδηγία MIFID θα μας βοηθήσει, αλλά χρειαζόμαστε εξουσίες για να μπορούμε να απαγορεύουμε κάποια προϊόντα ή κάποιες δραστηριότητες. Ε, κατ' εξαίρεση βέβαια, αλλά καλό θα είναι υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Και επίσης ε, θα πρέπει να σημειώσουμε κάποια πρόοδο και στα κίνητρα, γιατί έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις αποδοχές ε, στις επενδυτικές εταιρείε. Υπάρχει όμως και το θέμα των εναυσμάτων, των κινήτρων που δίνονται για τον ε, παραγό του προϊόντος απέναντι στον σύμβουλο που το προωθεί, που το προτείνει. Και αυτή η διαδικασία παροχής συμβολών ε, επηρεάζεται υπερβολικά από τα κίνητρα που δίνεται. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε ένα μοντέλο απλώς αποκάλυψης, αν τα αρχικά κίνητρα δεν είναι σωστά. Ναι. Και αν περάσουμε σε ένα μοντέλο πληροφόρησης, ε, θα είναι δύσκολο ε, για μας ως εποπτική αρχή να αντισταθμίσουμε τα κίνητρα εφόσον δεν είναι σωστά και δεν, δίνουν τα, δεν δίνονται τα σωστά κίνητρα για τη σωστή παροχή συμβουλών. Ευχαριστώ. Ανδρέα πολλές ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω έτσι σύντομα για την ομάδα ενδιαφερομένων. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε την ισορροπία και νομίζω ότι έχουμε μια διαφοροποιημένη σύνθεση. Ξέρω ότι κάποιοι ενδιαφερόμενοι, κάποιες ομάδες ενδιαφερομένων, οι καταναλωτές και τα συνδικάτα δεν είναι ευχαριστημένα. Ε, έβαλαν, έχουν διαβιβάσει παράπονα προς τον διαμεσολαβητή και περιμένουμε ο διαμεσολαβητής να κάνει την αξιολόγησή του και εν συνεχεία θα ξανασκεφτούμε το θέμα. Να τονίσω όμως ότι η ομάδα των ενδιαφερομένων δεν είναι το μόνο κανάλι για την αλληλεπίδραση με αυτές τις ομάδες. Έχουμε τακτικές συνεδριάσεις δύο φορές το χρόνο με αυτές τις ομάδες. Θέλουμε, τι? Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις τους. Και νομίζω ότι οι επαφές αυτές ε, εξελίσσονται πολύ ομαλά. Και όταν έχουμε και την απόφαση του διαμεσολαβητή θα δούμε ποια θα είναι η σύνθεση στο μέλλον της ομάδας ενδιαφερομένων. Πάντως ε, συγχαίρω την προσπάθεια της ομάδας αυτής, ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ε, είναι μια πολύ ε, καλά εκπροσωπημένη ομάδα κτλ. Τώρα για τις διαφορές και τις ομοιότητες. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Γκίκολτ για το πώς έθεσε το θέμα. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσέγγιση μας. Για τις υποχρέωσεις πληροφόρησης. Ξεκινάμε με μια πλατιά γκάμα, μιλάμε και απευθυνόμαστε και στα μικρά ιδρύματα και κατά τη διάρκεια της συζήτησης συνειδητοποίησαμε ότι επηρεάζονται ακόμα και οι μικρότερες τράπεζες. Και τώρα έχουμε ένα πρότυπο που θέλει να ε, εφαρμόσει αυτές τις υποχρεώσεις, ε, τις υποχρεώσεις δηλαδή πληροφόρησης για χρηματοπιστωτικά θέματα προς όλους. Είναι πολύ σημαντικό επίσης ε, να έχουμε μορφία γιατί υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις πληροφόρηση και με βάση την εθνική νομοθεσία για τους ε, χρηματοπιστωτικού ομίλου ομίλους με τερογενεί δραστηριότητες. Ε, θέλουμε να, να, να μεταρρυθμίσουμε εντελώ τους ομίλου αυτούς. Εγώ θέλω να πείσω τους ανθρώπους μου να κάνουν πραγματικά ριζική αναδιάρθρωση. Η οδηγία ε, για τους ομίλους θέλουμε να καταλάβουμε βοήθησε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το γεγονός ότι είχαμε αυτές τις ε, διατάξεις ε, μας βοήθησε με διατάξεις για τους ε, χρηματοπιστωτικούς ομίλους ή μήπω πρέπει να αλλάξουμε, τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε. Και βέβαια εν αναμονή της Τραπεζικής Ένωσης πρέπει να δούμε πραγματικά τι θα κάνουμε αυτό το νομοθέτημα. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν είναι αρκετά ισχυρή νομοθεσία για να αλλάξει πραγματικά τα πράγματα για, τις, για τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς ομίλους. Για την προστασία των καταναλωτών. Όπως σας είπα, δουλεύουμε πάνω στα ενυπόθεκα δάνεια, τον ενυπόθηκο δανεισμό και θα έχουμε σύντομα κατευθυντήρες γραμμές για την, τον υπεύθυνο δανεισμό με υποθήκες. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και για την κρίση που βιώνουμε θα πρέπει να δούμε πώ αλληλεπιδρούν οι τράπεζες με του καταναλωτές όταν οι καταναλωτές έχουν ε, δυσκολίε να αποπληρώσουν το δάνειό τους, το υπόθηκο δάνειο. Για το ETF, για τα κεφάλαια ε, που είναι συγμένα στο χρηματιστήριο, κάνουμε δουλειά, συντονιζόμαστε με την ΕΣΜΑ, ε, λαμβάνουμε υπόψη μας τον κίνδυνο και κάνουμε διαχείριση του κινδύνου. ασχολούμαστε με τους, ε, ερχόμαστε σε διάλογο με τους οργανισμούς ε, αυτών των κεφαλαίων, των ETF, των εισηγμένων στο χρηματιστήριο και θα ετοιμάσουμε μία έκθεση σύντομα για το Contacts for Difference και για τα διαφωμένα προϊόντα και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και την σκοπιά του καταναλωτή. Προσωπικά θεωρώ ότι πιέσαμε πολύ τις τράπεζες να συλλέξουν ε, κεφάλαιο και οι τράπεζες αντιμετώπισαν πάρα πολλές δυσκολίες στη χρηματοδότηση. Δηλαδή, εκεί που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την ισχύ τους, ούτω ώστε να μοιράσουν στους ιδιώτες επικίνδυνα προϊόντα, περίπλοκα προϊόντα χρηματοδότησης. Ε, επειδή ακριβώς αυτό είναι τεράστιο θέμα, θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα ε, στο Συμβούλιο των Εποπτικών Αρχών. Επίσης, τι παραθυράκια αφήνουμε ενδιαφέρον θέμα. Μας δώσατε σημαντικές αρμοδιότητες σε τομείς ε, της παραβίασης του δικαίου, στη μεσολάβηση, προστασία των καταναλωτών και στις έκτακτες ε, και κατεπίγουσες ε, καταστάσεις. Αυτές οι εξουσίες συνδέονται με την ύπαρξη ή όχι νομοθετημάτων. Ή μάλλον υπάρχουν νομοθετήματα. Ήταν δύσκολο να ενεργοποιήσουμε αυτές τις αρμοδιότητες, γιατί ας πούμε σκεφτείτε τις τράπεζες, εκεί δεν υπάρχει σχετικό κανονισμός. Ή, εν δεν έχουμε άμεσα εφαρμόσιμου κανόνε. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το θέμα, το θέμα με τα παραθυράκια και σε ορισμένες περιπτώσεις έχω την εντύπωση ότι ή έχουμε τρομερά ήπια εργαλεία ή προσπαθούμε να πείσουμε τις εθνικές αρχές να συνεργαστούν ή έχουμε ας πούμε τον μπαζούκα που τους πυροβολεί κατά κέφαλα με επίσημες διαδικασίες. Δηλαδή λείπει κάτι το ενδιάμεσο ανάμεσα στο τρομερά χαλαρό και στο τρομερά αυστηρό. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι η καλύτερη συνεισφορά στη συζήτηση, αλλά ε, σας το αφήνω να το σκεφτείτε. Επίσης, το θέμα της διακυβέρνησης. Ε, είμαστε σε φάση επιτροπής τώρα. Ε, για να περάσουμε και να γίνουμε πραγματική αρχή, πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα. Και κάποιες από τις ιδέες της Κομισιόν ε, για την ε, υλοποίηση της Τραπεζικής Ένωσης, την ε, αντίστροφη πλειοψηφία κτλ. Όλα αυτές τις ιδέες είναι ενδιαφέρουσες και πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω. Για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Θα ήθελα να σας πω ότι, ναι, καταρχήν, μόνο ένα ελάχιστο τμήμα ή μάλλον με τα τελικά νούμερα που έχουμε λάβει, Ξέρουμε ότι 107% της έλλειψης ε, καλύφθηκε με κεφαλαιακά μέτρα και το ποσοστό μείωσης ε, του δανεισμού είναι 0,8%. Είναι πολύ μικρό. Και το περισσότερο από αυτό το ζητάνε ε, οι κρατικές αρχές, απομόχλευση που ζητάνε οι κρατικές αρχές. Ε, αυτά που είπαμε εμεί με τη σύστασή μα δεν οδηγούν σε απομόχλευση. Παρ' όλα αυτά έχετε δίκιο. Συμβαίνει απομόχλευση και κυρίω συμβαίνει σε δύο τομεί. Καταρχά, στο leasing. Εκεί προχωρούν γρήγορα οι τράπεζε σε τέτοιου τομεί. Ε, στο global banking που προωθείται, εν πάση περιπτώσει, χάρη στο δολάριο, ε, το δεύτερο είναι η απομόχλευση σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το κρατικό τους χρέος. Οφείλεται και στη ζήτηση αυτή η απομόχλευση. Αλλά οφείλεται και στο ότι ο τραπεζικός τομέας, ο τραπεζικός κλάδος γίνεται πιο περιοριστικός θα έλεγα, πιο προσεκτικός ε, στο δανεισμό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, νομίζω πρέπει να απομοχλεύσουμε. Μπήκαμε στην κρίση με υψηλό επίπεδο μόχλευση, πρέπει να καταλήξουμε με, σε, χαμηλότερη μόχλευση. Υπάρχουν καλοί τρόποι απομόχλευση. Ε, η συγκέντρωση κεφαλαίου είναι ένα καλό τρόπο απομόχλευση. Η διάθεση ε, περιουσιακών στοιχείων σε τομείς ε, που δεν είναι κρίσιμοι ας πούμε, επιχειρηματικά ε, είναι ένας άλλος καλός τρόπος. Η μείωση της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, η αναγνώριση των ζημιών είναι πολύ καλός τρόπος απομόχλευσης. Ίσως δεν έχει γίνει 100% όπως θα έπρεπε. Η μείωση όμως του δανεισμού είναι κακός τρόπος απομόχλευσης. Ε, ο τρόπος νομίζω που διαμορφώσαμε και διατυπώσαμε την ε, σύστασή μας θα μας βοηθήσει να κάνουμε μια εξισορρόπηση. Για το δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στείλαμε μια ε, έκθεση στην Κομισιόν με κάποιες ιδέες για το τι μπορεί να γίνουν και τη, στείλουμε και, τη στείλαμε και στην Επιτροπή σας και είμαστε έτοιμοι να τη συζητήσουμε. Με δύο λόγια, ποια είναι η άποψή μας. Ίσως είναι επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την, το δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω στάθμισης, του κινδύνου των τραπεζών. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά σε περίοδο, περίοδο ύφεση, θα πρέπει να έχουμε ελάφρυνση του κεφαλιακού βάρους που μπορεί να απαιτηθεί όταν τελειώσει η κρίση. Ξέρετε πολύ καλά, αν έχουμε ύφεση, δυσκολεύει ο δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και εκεί είναι που πρέπει να παρέμβουμε. Έμα, εσεί έχετε όλε τι ωραίε ερωτήσει. Λοιπόν, Γκαμπριέλ. Ναι, θα προσπαθήσω και εγώ να καλύψω τα, τα βασικά για τι ομάδε των ενδιαφέρομενων και ευχαριστώ, Σβέν, για την ερώτηση. Νομίζω πω οι συνάδελφοί μου ήδη απάντησαν. Από τη δική μα την πλευρά προσπαθήσαμε να ε, έχουμε βεβαίω ε, ισορροπημένη σύνθεση και ποιότητα βεβαίω των ανθρώπων εκεί πέρα που μας συμβουλεύουν. Επίσης, κάτι άλλο που έχει σημασία είναι το επίπεδο των ε, πόρων που δεν έχουν βεβαίως οι ομάδες των καταναλωτών. Από τη μεριά του κλάδου έχουν, προετοιμάζονται κτλ. Ε, από την πλευρά των καταναλωτών είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό το οποίο κάνουμε και συμφωνήσαμε τους εκπροσώπους των καταναλωτών και ενδιαφερομένων παραδείγματο χάρη στις ασφάλειες είναι για τη δικιά μας τη δουλειά και τις πρωτοβουλίες μας έχουμε ετοιμάσει κάποιες βασικές σημειώσεις, κάποια γεγονότα, παραδείγματος χάρη το τι είναι η οδηγία για τη φερικαιότητα 2 για να μπορέσουν να έρθουν στη συζήτηση πιο προετοιμασμένοι από πλευράς καταναλωτών για να βοηθήσουμε και τις ομάδες των ενδιαφερομένων για να έχουμε μια καλή συζήτηση. Νομίζω πως είμαστε ικανοποιημένοι με τη συνεργασία που έχουμε. Για το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης και των χρηματοασφαλιστικών ομίλων. Νομίζω πως πρέπει να αντιληφθούμε ξεκάθαρα το τι πρέπει να γίνει με το θέμα των ομίλων. Αυτό το οποίο προσπαθούσα να εξηγήσω είναι πως είναι γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί ε, απευθείας να έχει αρμοδιότητα για τις ασφαλιστικές εταιρείε, ε, αυτό το αναφέρει η συνθήκη, μπορεί να υπάρξει μια συμπληρωματική υποπτία στο επίπεδο των ομίλων, οπότε δεν έχει άμεσες αρμοδιότητες ε, μόνο στο επίπεδο της μητρική εταιρεία χαρτοφυλακίου, αλλά βεβαίω συχνά η μητρική εταιρεία χαρτοφυλακίου είναι ασφαλιστική εταιρεία και δεν ξέρω μετά πώ ε, μπορεί να έχει τέτοιε αρμοδιότητε. Όπω είπα, Σημαντικό είναι να το δούμε και από τη σκοπιά των, ασφαλιστικών εταιριών. Και μπορεί να γίνουν κάποια βήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. όσον αφορά τα εσωτερικά α, μοντέλα. Α, περνάμε τώρα στη φερεγγιότητα 2 για εσωτερικά μοντέλα για τα κεφάλαια. Βλέπουμε ήδη δυσκολίες ε, στην προσέγγιση μεταξύ των διαφόρων αρχών όσον αφορά την περίοδο πρώτων ετήσεων. Εγώ θεωρώ πως θα πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στην ΕΙΟΠΑ για να υπάρχει μία συνοχή σε αυτά τα εσωτερικά μοντέλα και βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει και στο πλαίσιο των ομίλων στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης να είμαστε και εμείς συνομιλητές ε, της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας. Στο μέλλον τώρα αν υπάρχουν στοιχεία μπορούν να βελτιωθούν. Παραδείγματο χάρη ε, πρόσβαση σε ατομικά δεδομένα. Ναι, έχουμε τέτοια πρόσβαση σε κάποιες ε, περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να είναι αυστηρές οι εθνικές εποπτικές αρχές. Εγώ παραδείγματο χάρη θα καλωσόριζα κάτι πιο ξεκάθαρο στην αναθεώρηση των κανονισμών σε σχέση παραδείγματο χάρη με τι ποιοτικέ μελέτες επιπτώσεων όσον αφορά ατομικά στοιχεία που μεταδίδονται στην ΕΙΟΠΑ, γιατί βεβαίως θα χρειαζόμαστε και αυτά. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στο μέλλον, όταν θα κάνουμε τη δική μας ανάλυση, τις δικές μας έρευνες, να πάμε απευθείας στις ασφαλιστικές εταιρείες και να κάνουμε απευθείας μαζί τους διάλογο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί. Όπως ανέφερα στην αρχή για την προστασία των καταναλωτών και τις αρμοδιότητες του άρθρου 9, αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό γιατί αν δεν υπάρχει στη βασική νομοθεσία η δυνατότητα να δράσουμε, να περιορίσουμε προϊόντα, υπάρχουν κάποιες ε, προσδοκίες ε, βεβαίως που έχει δημιουργήσει η ρυθμιστική αρχή, εσείς τα έχετε βάλει στο άρθρο 9, που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε όμως χωρίς ε, αυτές τις αλλαγές στην οδηγία, στην νομοθεσία. Και Κάτι άλλο το οποίο μπορεί οπωσδήποτε να βελτιωθεί αφορά την πλευρά των συντάξεων στον τρίτο πυλώνα, στα ατομικά προϊόντα όπου δεν υπάρχει ευρωπαϊκή προσέγγιση. Νομίζω πως οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια, να ε, υπάρξει αυτή η οικοδόμηση του οικοδομήματο τη κοινωνική ασφάλεια στην Ευρώπη και βεβαίω αυτέ τι τάσει κάνουμε και στην Κομισιόν. Για τη Φεργιώτα 2 τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι η δική μου ευθύνη η, εφαρμογή. Αυτό το οποίο μπορώ οπωσδήποτε να πω είναι πως καλό είναι Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα στείλει ένα μήνυμα προς τα έξω πώς θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Και βέβαια γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά το πακέτο αυτό των μακροπρόθεσμων εγγυήσεων και προϊόντων. Εμείς ε, ευπρόσδεκτη βλέπουμε αυτή την ευθύνη για να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση και να, κάνουμε, να σας στείλουμε τα αποτελέσματα. Θα το κάνουμε αυτό, με τρόπο ανεξαρτό, αλλά πρέπει να είναι και σαφές. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε προς τα πίσω, αυτό είναι σαφές. Η φερικαιότητα 1 που ισχύει τώρα, και θα σας τα πω ξεκάθαρα, δεν καλύπτει τους κινδύνους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το έχετε στα χέρια σας, ε, έχετε τα πίνακες κινδύνου που φτιάχνουμε εμείς. Εάν δείτε τους κινδύνους εδώ πέρα που υπάρχουν, ε, οι περισσότεροι από αυτούς που αυτή ε, τη στιγμή διατρέχουμε δεν καλύπτονται από τι κεφαλαϊκέ απαιτήσει τη φερεγκαιότητα 1. Είναι θεμελιώδε λοιπόν το ζήτημα. Πρέπει να εφαρμοστεί η φερεγγιότητα 2. Χρειάζεται ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα και μια λύση αξιόπιστη. Γιατί και στο διεθνέ επίπεδο έχει σημασία αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και προ τα έξω. Όσον αφορά τώρα το πώς μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία ασφαλιστικές εταιρείε ε, και συνταξιδοτικά ταμεία. Ναι και αυτό έχει σημασία. Πρέπει συνταξιδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείε να επενδύουν μακροπρόθεσμα. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουν υπό ένα υγιέ ρυθμιστικό περιβάλλον. Το χειρότερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για τη χρηματοδότηση της οικονομία είναι να υπάρχει αίσθηση πω μειώνοντα τι απαιτήσει ε, σε ασφαλιστικές ε, εταιρείες και στα τα ταμεία, βοηθούμε την ανάπτυξη. Το έχουμε δει αυτό που έχει οδηγήσει σε άλλου τομεί. Χρειαζόμαστε βιώσιμη ανάπτυξη. Βιώσιμη θα είναι μόνο εάν έχουμε υγιεί ρυθμιστικέ ε, απαιτήσει για τι εταιρείε ε, στον τομέα. Και βεβαίω ε, οι εταιρείε αυτέ και τα ταμεία οπωσδήποτε θα βοηθήσουν τη χρηματοδότηση της οικονομίας και χρηματοδότηση έργων, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, οπωσδήποτε είναι ένας τομέας ε, που θα μας απασχολήσει. Αλλά ας μην προκαλέσουμε, σας παρακαλώ, περισσότερους κινδύνους και μεγαλύτερες κρίσεις. Ας διδαχτούμε από αυτή την κρίση. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες ε, ήταν ε, και μακροσκελής οι ερωτήσεις. Έχουμε δύο κομιγύρους τριών ομιλητών. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Πίτερ Σκίνερ, Ιβό και Δεκί Φόρτ. Ευχαριστώ, θα είμαι λακωνικός για την εξοεδαφικότητα. Δεν είναι και πολύ αστείο θέμα. Πιστεύετε ότι καλύτερα να την καλύψουμε με εξάντε ή εξπόστη νομοθεσία. Τι γίνεται, ποια είναι η την νομοθεσια τι γινεται ποια λύση. Για την χρηματοδότηση είπατε, είτε 100% κοινοτική χρηματοδότηση ή μια εισφορά από τον κλάδο και το προτιμάτε. Και πώς θα το χρησιμοποιήσετε όμως ε, σε σχέση με την μεικτή Επιτροπή, κάτι που δεν αναφέρθηκε. Και για τις συντάξεις, ε, για τον Καμπριέλ της ΕΙΟΠΑ. Διάβασα στην ιστοσελίδα ότι δεν θα ε, διευρύνεται το πεδίο. Αναφερθήκατε και σε ατομικές συντάξεις. Συμφωνώ πάντως για τη Θεργιώτα 2, Όντως, μερικοί θα προτιμούσαν ε, την εφαιρεγγιότητα 1 ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, αλλά ε, δεν συμφωνούμε με κάτι τέτοιο και ελπίζουμε να εφαρμοστεί δύο. Ο Ήβο. Μία ερώτηση για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, τον κύριο Νηρία. Κύριε Πρόεδρε, δεδομένες της νέας πρόταση για την ενιαία τραπεζική εποπτεία μαζί με την ΕΚΤ. Η νέα τραπεζική αρχή θα είναι αρμόδια για τον ορισμό και την εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις τράπεζες για τις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι η δική σας θέση, πώς πιστεύετε ότι η διαδικασία λήψη αποφάσεων στην ΕΤΑ δεν θα παραγωνίσει τα μέλη που δεν ανήκουν στην Ελληνική Ένωση και δεν θα έρθουν σε δυσμενή θέση σε σχέση με τα μέλη που θα είναι κράτη, που θα είναι μέλη και της Τραπεζικής Ένωσης. Η Βίκη. Έχω ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Χαίρομαι για την πρότασή σας για αυστηρούς κανόνες για ρευστότητα του κεφαλαίου, γιατί Ακούω συνέχεια την Επιτροπή ε, που λέει θα εφαρμόσουμε τη Διεθνή Συμφωνία της Βασιλείας και στην Ευρώπη. Ναι, και πιστεύω ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τα παθήματα του παρελθόντος και να προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού να εφαρμόσουμε διεθνεί συμφωνίες για τη ρευστότητα του κεφαλαίου. Θεωρείτε ότι θα έχουμε ένα, μία δέσμη κανόνων για την Ευρωζώνη και χαλαρότερους κανόνες ε, για τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα ήταν απαράδεκτο. Και ε, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το CRR, αν δούμε το κείμενο του Συμβουλίου για, το κεφαλαί... για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Θα έχουμε συμμόρφωση με τη Βασιλεία για το κεφάλαιο. Μιλήσατε για διαφορά 300 μονάδων βάσης. Συνάδει με τη Βασιλεία, με τη Συμφωνία της Βασιλείας. Και και θα έχει διαφορά αν οι μεγάλες τράπεζες συμμορφωθούν και οι μικρές όχι. Ποια θα είναι η διαφορά. Τώρα ως προς τη ρευστότητα. Έχουμε τη νέα εκδοχή της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ρευστότητα. Ε, πώς θα βάλετε στο, δρόμο τους, αυτούς τους λόγους ρευστότητας. Γιατί φαίνεται ότι τα διέγραψε όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το παράρτημα και το μεταβιβάσιμο πριν το στοιχείο του ενεργητικού. Συνεννοήθηκε μαζί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν υποβάλει τις νέες της προτάσεις. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση που κάνατε, την αξιολόγηση για, την, για το δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα ληφθεί υπόψη στη νέα οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις και το CRR. Θα το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μας ε, αυτό που προέχει είναι η ανεξαρτησία σας ε, και ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων. Και ε, πώς θα εξασφαλίσετε τη διατήρηση αυτής της ανεξαρτησίας αν κάποιος επόπτης ελέγχει την πλειοψηφία των ψήφων ή σχεδόν την ειδική πλειοψηφία των ψήφων. Αν τα καταφέρετε να περιοριστείτε στο πεντάλεπτο καθένας, ίσως ολοκληρώσουμε εγκαίρως και τον τρίτο κύκλο. Θα ήθελα να, να ξεκινήσω με το θέμα της εξοδαφικότητας. Η εξοδαφικότητα α, σχετίζεται και με την αλληλεπίδραση των χρηματαγορών. Και το, αδύναμο, και το βασικό στοιχείο της εξοδαφικότητας είναι ε, το αδύναμο στοιχείο είναι δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν συνθήκες ε, ίσου ανταγωνισμού. Οπότε ε, έξω δραστηριότητες, επιχειρήσεις που παρέχουν δραστηριότητες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δεσμεύονται από τις συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Γιατί θα πρέπει οι προδιαγραφές και πρότυπα να ισχύουν και για τις δοκινοτικές και για τις εξοκοινοτικές επιχειρήσεις. Ένα είδος εξοδαφικότητας βέβαια είναι αναπόφευκτος ό,τι αφορά τις αλληλοεπιδρόμενες αγορές. Νομίζω ότι το ίδιο κάνει και η Ευρώπη. Όταν έχουμε μια, ε, ένα fund manager που έρχεται ε, από εξωκοινωτική χώρα εντός της ε, Ευρώπης, σε επιβάλλουμε ίδια πρότυπα με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαχείριση εναλλακτικών ταμείων. Τώρα, όταν, και, όταν αρχίζουμε και έχουμε διαφορές στην εποπτεία, επειδή υπάρχει διαχωρισμός των συστημάτων, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το συντονισμό εντός του G20 και ένα άλλο πρόβλημα στο τομέα του κανονισμού ΕΜΙΡ είναι ότι όταν ε, θεωρούμε ότι ένα σύστημα τρίτης χώρας είναι ισοδύναμο με το ευρωπαϊκό, ε, στηριζόμαστε σε αυτό. Βέβαια αυτή η συζήτηση είναι πολύ δύσκολη και για τον κανονισμό ΕΜΗΡ, για τις υποδομές της αγοράς. Έχουμε άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δούμε τι γίνεται με το CC και SDC. Δεν θέλουμε να γιατί λένε δεν θέλουμε να στηριχθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία ή να στηριχθούμε λιγότερο σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και το πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι όχι μόνο ε, ότι υπόκειται στην ευρωπαϊκή ε, εποπτεία από τι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, αλλά υπόκειται και στην αμερικανική εποπτεία. Και εργαζόμαστε σκληρά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προωθήσουμε αυτό το μοντέλο Έχουμε την υποστήριξη των συναδέλφων από την Ασία, γιατί οι Ασιάτες προτιμούν αυτό το μοντέλο της αμοιβαία αναγνώρισης, αλλά είναι δύσκολο να, πολύ πιο δύσκολο να πείσουμε τους Αμερικανούς συνομιλητές μας. Πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε και ήδη διαπιστώσαμε κάποια πρόοδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. ή θέλουμε πλήρω κοινοτική χρηματοδότηση καθόλου χρηματοδότηση δηλαδή από τις εθνικές αρχές. Και αυτό είναι ο απότερο σκοπός μας. Ίσως τελικά προκριθεί ένας συνδυασμό με κάτι, ένα τμήμα που προέρχεται από τη βιομηχανία, από τον κλάδο και ένα από την από το κοινοτικό προπολογισμό. Τώρα συγκεντρώνουμε τα ε, κονδύλια από τις, ε, τους οίκους ε, αξιολόγηση. Το ίδιο θα κάνουμε και με τα εμπορικά μητρώα, τα μητρώα συναλλαγών μάλλον. Ίσως εφαρμοστεί μία εισφορά από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τώρα, για την ανεξαρτησία. Θα πρέπει να υπάρχει νομική βάση για την επιβολή αυτής της εισφοράς. Τώρα, αυτή η εισφορά μειώνει την ανεξαρτησία. Ήμουν και στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή με 80% χρηματοδότηση από την αγορά και 20% από την ε, κυβέρνηση. Θα πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες φορολογίας και οι εξουσίες. Ε, δεν έχω ε, ανησυχίες για την ανεξαρτησία. Θα πρέπει να εντοπίζουμε τους, α, ε, τους συμμετέχοντες στην αγορά και να ξέρουμε από ποιους θα συλλέω, θα συγκεντρώνουμε αυτά τα κονδύλια αυτές τις φορές. Αντρέα, πάλι εσένα σου έτυχαν οι καλέ ερωτήσει, αλλά δεν έχει τόσο χρόνο όσο την άλλη φορά. Ναι, για το πρώτο ερώτημα για τη λήψη αποφάσεων και το που βρίσκονται ενώπιον της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Κοιτάξτε, το άρθρο 42 του καταστατικού μας λέει πως όσοι είναι στο δουσού μας πρέπει να εργάζονται προς το ευρωπαϊκό συμφέρον και να μην λαμβάνουν οδηγίες ή να ζητούν ε, συμβουλές από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς και μετά ψηφίζουμε με ειδική πλειοψηφία, οπότε έχουμε κάποια εθνική αντιπροσώπευση, εάν θέλετε, κάτι το οποίο δημιουργεί ένταση. Κατά την άποψή μου, η ιδέα της Κομισιόν να πάμε σε ανεξάρτητα πάνελ σε κάποιους ε, τομείς που θα λαμβάνουν δηλαδή τεχνικές αποφάσεις και όχι πολιτικό παζάρι, πάνελ ειδικών που θα σχεδιάζουν ε, ε, κάποιες ε, προδιαγραφές ε, και θα ψηφίζουμε κάποιες αντίστροφες τηλεοψηφίες, νομίζω είναι κάτι που αξίζει να ερευνήσουμε. Και έτσι θα αποφευχθεί νομίζω το ότι οποιαδήποτε μία εποπτική αρχή ή συμμαχία εποπτικών αρχών θα μπορούσαν να περάσουν τις απόψεις τους. Αυτή είναι η απόψή μου και νομίζω πως η Κομισιόν έχει κάνει το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα και τη συμμόρφωση. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή της Βασιλείας κάνει μία αξιολόγηση με μία διαδικασία από ομότιμους, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πράγματι κάποιοι τομείς στους οποίους το κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλίνει από αυτό της Βασιλείας και υπάρχουν καλοί λόγοι γιατί αφενός εφαρμόζουμε τους κανόνες σε 8.000 ε, τόσες ε, τράπεζες, ενώ σε άλλες χώρες ε, αυτά ισχύουν μόνο για τις μεγάλες και διεθνείς τράπεζες. Από την άλλη, νομίζω πως πρέπει να αναρωτηθούμε, κυρίως όσον αφορά το κεφάλαιο, το κεφάλαιο είναι η βασική μου ανησυχία. Ε, ενώ αντιλαμβάνομαι βεβαίως πως θα πρέπει ίσως να προσαρμόσουμε τις απαιτήσει σε αυτά τα οποία ζητάνε οι συνεταιριστικές τράπεζες οπωσδήποτε, αλλά όλα τα μέσα θα πρέπει να είναι εξίσου ε, στεναρά και όσον αφορά την απορρόφηση ζημιών και την ευελιξία κτλ. Και όσο λιγότερα ευελιξία υπάρχει τόσο το καλύτερο. Εγώ θα στήριζα, το είπα ήδη και την προηγούμενη φορά, πως ε, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα πρέπει να μπορεί να επιτηρεί την ποιότητα των κεφαλαίων μέσων. Όσον αφορά τη ρευστότητα, ναι, η κατάσταση είναι κάπως διαφορετική. Εντάξει, η Κομισιόν ε, συνεργάζεται καλά μαζί μας, ε, γεγονός είναι αυτό. Όσον αφορά τη ρευστότητα λοιπόν υπάρχει μια λεπτή ισορροπία που πρέπει να βρεθεί. Αφενός χρειάζονται ισχυρέ και απαιτήσει ρευστότητα για να αλλάξουν επιχειρηματικό μοντέλο οι τράπεζε. Πρέπει να γίνει αυτό. Από την άλλη πρέπει να αποφύγουμε το να σκοτώσουμε έτσι την ε, διατραπεζική αγορά που έχει φτάσει πολύ κοντά σε αυτό το σημείο και κάνουμε κάποιες ε, σκέψεις στο διεθνές ε, επίπεδο και θα χρειαστεί νομίζω λίγο περισσότερος χρόνος. Θα κάνουμε μια έκθεση του χρόνου εάν η νομοθεσία εξακολουθήσει να έχει αυτές τις απαιτήσεις. Ήδη συλλέγουμε στοιχεία από διάφορες τράπεζες και έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε στοιχεία από όλες τις τράπεζες για να έρθουμε σε εσά με προτάσεις για το τι πρέπει να κάνουμε για το, τον λόγο ρευστότητας, για την εξαρτησία νομίζω αναφέρθηκα ήδη. Οπότε θα σταματήσω εδώ. Μάλιστα. Εμείς θα θέλαμε να το διαπραγματευτούμε τις ερχόμενες εβδομάδες, όχι του χρόνου η ερμηνεία μου είναι πως η Κομισιόν διέγραψε τις απαιτήσει να αναφέρονται κάποιοι σε εσά, όχι να αναφέρονται πράγματα δημόσια, αλλά σε εσά, ε, τη ρυθμιστική, ε, την εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές που έγιναν. Κοιτάξτε, για εμένα το ζήτημα είναι να διασφαλίσουμε πως θα έχουμε στην ε, νομοθεσία μία εντολή στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να εκδίδει τεχνικές προδιαγραφές για τη συλλογή δεδομένων στην ενδιάμεση φάση. Δεν μιλάμε βεβαίω θα γίνει στη φάση της μελέτης, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν πρώτα απ' όλα οι απαιτήσει πριν ε, καταλήξουμε σε κάποιες ε, στην έκθεση των μονίμων απαιτήσεων και ελπίζω να είναι αρκετά ευρία η εντολή για να μας επιτρέψει να συλλέξουμε πληροφορίες ε, σε ένα αρκετά μεγάλο φάσμα μέσων για να καλύψουμε σωστά τις απαιτήσει. Έχουμε ήδη όμως ε, πει στον κλάδο πως ε, θέλουν, υπάρχουν κάποια μέσα που θέλουμε να συμπεριληφθούν όπως ε, μετοχικό κεφάλαιο ή αξιόγραφα τα οποία βασίζονται σε στεγαστικά δάνεια κτλ. Τα οποία κατά την άποψή μα δεν είναι καθόλου αξιόπιστα. Φυσικά θέλουμε γενικούς κανόνες για την ε, εξοδαφικότητα και στις ασφαλιστικές εταιρείε και στην ΕΙΟΠΑ. Ε, υπάρχει η Εκτελεστική Επιτροπή που θέλει να υπάρχει μια ε, ευρωπαϊκή θεώρηση, ούτω ώστε να υπάρχουν πιο παγκόσμια πρότυπα για τις ασφαλιστικές εταιρείε. Αυτά ήταν η ιδανική λύση. Διαμέσως βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της προστασίας των καταναλωτών ε, και των ε, προστασία των εταιριών στην Ευρώπη. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ισοδυναμία, ούτω ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματική εποπτεία γενικά. Και, να, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να μπορούμε να βασιζόμαστε στα συστήματα των τρίτων χωρών. Αυτές τις αξιολογήσεις ισοτιμίας τις κάνουμε με την Ελβετία, με την Ιαπωνία, ε, έχουμε τελειώσει. Ετοιμάζουμε τις ε, ισοδυναμίες με 8 άλλες χώρες. Κοιτάμε τι στοιχεία κοινά έχουμε και έχουμε ξεκινήσει και την, ε, το εγχείρημα αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να δούμε τι κοινά έχουμε, τι διαφορές έχουμε. Θα κάνουμε διαβουλεύσεις ε, για αυτά τα θέματα των κοινών στοιχείων και των διαφορών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτόν τον τομέα ε, ελέγχουμε το θέμα. Φυσικά η τελική λύση θα ήταν να έχουμε παγκόσμια πρότυπα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και νομίζω ότι οι εποπτικές ε, αρχές των ασφαλιστικών εταιρειών πρέπει να το κάνουν αυτό. Για το θέμα της χρηματοδότησης και το, τη χρηματοδότηση 100% ή χρηματοδότηση μέσω εισφοράς. Εγώ θα ήθελα 100% χρηματοδότηση, αν γινότανε. Αλλά καθώς περνάει ο χρόνος και καθώς θα προχωράμε βαθμιδών, θα πρέπει τελικά να σκεφτούμε αν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες ε, εξουσίες άμεσης εποπτείας στις εποπτικές αρχές. Ε, και αυτό να το συνδυάσουμε με κάποιο τέλος, κάποια εισφορά. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα αμφισβητείται η ανεξαρτησία μας, η ανεξαρτησία τους. πάει χέρι με χέρι με τις περισσότερες εξουσίες που θέλουμε να δώσουμε σε εποπτικές αρχές. Τώρα, για τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Έχουμε στείλει τις συμβουλές μας στην Κομισιόν για αναδιάρθρωση της σχετικής οδηγίας ε, για πρώτη φορά θα συλλέξουμε τώρα δεδομένα από τα διάφορα συνταξιωτικά ταμεία στην Ευρώπη. Θα το κάνουμε το δεύτερο εξάμεινο του 2012 και είναι πολύ σημαντική η διαδικασία για την αξιολόγηση των ιδεών μας και προτάσεών μας, ούτως ώστε να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες των συνταξιωτικών ταμείων στις διάφορες χώρες. Μπορούν να ενταχθούν ε, σε αυτό το συνολικό πλαίσιο. Πόσο πρακτικό είναι αυτό. Πώς μπορούμε να το διαφοροποιήσουμε, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη υποπτή ανάλογη με τον ε, κίνδυνο παρουσιάσουν τα συνταξιωτικά ταμεία. Γιατί σα το πω ανοιχτά. Και τα συνταξιωτικά ταμεία ε, θα πρέπει να κάνουμε τεστ αντοχή. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι όλα πάνε καλά, γιατί δεν είναι. Υπάρχουν κίνδυνοι και εκεί. Έχουμε αυτό το σενάριο χαμηλών επιτοκίων που σκοτώνει τα συνταξιωτικά ταμεία. Και υπάρχουν δύο στάσεις. Ή θα συνεχίσεις να στρούθω μιλίζει και να θεωρεί ότι όλα είναι καλά και θα το αντιμετωπίσεις αργότερα βέβαια. Στο μέλλον θα το βρει μπροστά σου ή θα προσπαθήσει να κάνει ένα τεστ με ανοιχτά τα μάτια. Φυσικά, όταν είμαστε πιο διαφανείς, όταν κάνουμε υπολογισμού των κινδύνων, δεν σημαίνει ότι ντε και καλά πρέπει να κάνουμε αμέσω ανακεφαλαιοποίηση αυτών των ταμείων. Σημαίνει ότι και οι εργοδότε και οι εργαζόμενοι απλώ θα έχουν πιο καθαρή εικόνα για του κινδύνου και ποιο επομίζεται αυτού του κινδύνου. Και μετά ε, θα υπάρχει το κίνητρο για να ληφθούν μέτρα και αποφάσει. Πρέπει να το πούμε αυτό. Σε ορισμένε περιπτώσει τα ε, συνταξιωτικά ταμεία υπόσχονται συντάξει εργασία, απασχόληση α πούμε, ε, εντελώ ε, ανέφικτε. Είναι ευθύνη μου να το πω αυτό. Και το λέω πραγματικά με τα λόγου γνώσεως. Το έχω ξαναπεί αν διαβάσετε αυτά όσα έχω γράψει. Επίσης πρέπει να κάνουμε ε, μια ρεαλιστική δοκιμή είναι, των ταμείων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει στην Ευρώπη. Και οι τελευταίοι τρεις ομιλητές. Όλα Αντολίν και υποφαινόμενοι. Όλε. Ευχαριστώ. Οι διαπραγματεύσει ε, για τον επόμενο προπολογισμό, το προπολογισμό τη επόμενη χρονιά, ε, ε, έδειξαν μεγάλη διάσταση απόψεων ω προ τη... ως τους πόρους που θα πρέπει να αφιερωθούν στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Εμείς στην Επιτροπή μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο προπολογισμό των εποπτικών αρχών. Οπωσδήποτε. Συμβούλιο όμως και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν περικοπές σε πολλούς τομείς. Οπότε θα ήθελα να θέσω μια γενική ερώτηση. Το Συμβούλιο πρότεινε περικοπέ, Αν τελικά ε, εγκριθούν και γίνουν πραγματικότητα, ποιε θα είναι οι συνέπειε του, στις δικέ σα δραστηριότητε, Τι δυνατότητα πια θα έχετε να ανταπεξέλθετε στι ε, υποχρεώσει σα και στην ε, εντολή σα. Θα πρέπει να μειώσετε τι προδιαγραφέ, να υποβαθμίσετε το έργο σα ποια θα είναι οι συνέπειε των προτινόμενων περικοπών. Μα είπατε ποιε είναι οι ανάγκε σα ω προ τον προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πολύ χαμηλότερα κονδύλια από αυτά που είχαμε εμείς ε, προτείνει. Πώς βλέπετε την παρούσα κατάσταση, ποιες είναι οι πραγματικές σας ε, χρηματοδοτικές ανάγκες. Ε, θεωρείτε ότι είναι η ίδια κατάσταση με αυτή που επικρατούσε την Άνοιξη, υπήρξαν αλλαγές και αν ναι, γιατί και πού. Ο Αντολίν. Ευχαριστώ δύο ερωτήσει: μία για την δημοσιονομική σταθερότητα και η δεύτερη για τους καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, πώς θα βοηθήσετε τις χώρες που είτε έχουν υπαχθεί σε συστήματα διάσωση είτε χρηματοπιστωτικής ε, στήριξη. και σε ό,τι αφορά τους καταναλωτές. Έχουμε τις προτιμησιακές συμμετοχές στην Ισπανία. Είναι προϊόντα πολύ περίπλοκα, υψηλού κινδύνου, που τέθηκαν σε εμπορία ε, και αγοράστηκαν ακόμη και από μικρούς επενδυτές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες ε, αντιδικίες ε, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Να δοθούν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές Έχουμε τεράστιο πρόβλημα στην Ισπανία, οπότε είναι ρυθμιστικό πια το επίπεδο στο οποίο θα πρέπει να επιληθεί και όχι περιπτωσιολογικό. Σε ό,τι αφορά τι υποθήκε, έχουμε τριμερή διάλογο Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την οδηγία για τι υποθήκε. Αναφερθήκατε σε καταθετήριε γραμμέ. Φαντάζομαι θα συνοδεύσουν αυτή την πρόταση κοινοτική οδηγία. Έχετε κάποιε προβλέψει για το θέμα αυτών των υποθηκών. Μας ενδιαφέρει σε τι φάση βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές ε, ενέργειες. Σε ό,τι αφορά την ΕΙΟΠΑ, την περασμένη, το περασμένο Σεπτέμβριο είχατε υποβάλει μια έκθεση για την ε, χρηματοπιστωτική παιδεία ε, στα κράτη-μέλη. Έχετε νέα στοιχεία, θα ήταν πολύ χρήσιμα. Και η Πρόεδρος. Λοιπόν, σειρά μου τώρα. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις για την Τραπεζική Ένωση και την Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων που είναι πολύ σημαντική για μας αυτή τη στιγμή. Οπότε, Ανδρέα, αυτό το οποίο με ανησυχεί και ήσουν και εσύ στη συνάντηση εκείνη του ΕΚΟΦΗΝ είναι πως εάν δεν υπάρχει φρένο στην Τραπεζική Ένωση γιατί ξεκινάμε με ενιαία εποπτική αρχή και γίνεται εποπτική αρχή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τότε πως κόβεται ο δεσμός με τα κράτη και το δημόσιο χρέος, γιατί βεβαίως το φρένο θα μπει σε, κάποια, σε κάποιο επόμενο νομοθέτημα, οπότε έχουμε μια νομοθεσία που δίνει εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενώ ακόμα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ε, την ε, στηρίζουν και βρίσκονται από πίσω της και πολλά κράτη-μέλη λένε πως τα κοινοβούλια μας θα θέλουν να εμπλακούν. Και να πάω να βήμα παραπέρα. Αν το φρένο τελικά είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, αν πρέπει να συμπληρωθεί με λεφτά θα πρέπει ε, και εκεί πέρα θα θέλουν τα εθνικά κοινοβούλια να εμπλακούν και μετά το σύνολο των διαθέσιμων ε, ποσών σε ESM και FSF είναι το, της τάξης μεγέθους που διέθεσε το Ηνωμένο Βασίλειο στις ε, τράπεζές του στην κρίση. Οπότε, εάν έχουμε άλλη μια αισθημική κρίση, θεός φυλάξει, δεν θα επαρκούν νομίζω ε, αυτοί οι μηχανισμοί ασφαλείας. Πώς Κόβεται λοιπόν έτσι η σχέση αυτή την οποία αναφέρατε. ό,τι και αν κάνουμε οπωσδήποτε θα διαταράξει την έννοια αγορά. Εγώ θέλω να ξέρω πως τουλάχιστον θα ωφεληθούμε. Γιατί αλλιώς λέμε πως ωφελούμαστε σε κάτι και εντωμεταξύ έχουμε καταστρέψει κομμάτι της εσωτερικής αγοράς. Αυτό με ανησυχεί. Το άλλο θέμα το οποίο ρωτήσατε ή αναφέρατε ήταν αφορούσε την, ε, την ευελιξία. Και εδώ πέρα, συμφωνώ με την Βίκη, δεν είναι εδώ πέρα ε, εκτός Ευρωζώνης το κομμάτι όπου υπάρχουν ε, χαλαρές προδιαγραφές. Αλλά τι θα κάνουμε με, την μακροπροληπτική, με τις μακροπροληπτικές διαφορές που υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν φούσκες ε, στα ακίνητα στην Ιρλανδία, στην Ισπανία. Αυτό δεν θα εξαφανιστεί γιατί έχουμε μία, ε, μία νομισματική πολιτική. Εγώ κάθομαι εδώ πέρα με τον Γκέι Μίτσελ εδώ και 7 χρόνια και ρωτούσαμε τον ε, Τρισέ στο νομισματικό διάλογο τι θα κάνουμε για τη φούσκα των ακινήτων και για το ότι δεν ταιριάζουν τα επιτόκια στην Ιρλανδία. Αυτό δεν θα εξαφανιστεί από την μια μέρα στην άλλη. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Θα είναι οι εθνικέ εποπτικές αρχές αυτές οι οποίες θα δίνουν συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή πώ θεωρείτε ότι θα το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα, θα το σταματήσω αυτό τώρα το κομμάτι. Λοιπόν, για τη ρευστότητα θέλω να ακούσω την άποψη της ΕΣΜΑ, γιατί εγώ θεωρώ πως έχουν κλείσει οι ε, αγορές ε, χρημάτων γιατί έχουν τρομάξει και δεν ξέρουν τι συμβαίνει στις τράπεζες και οι επενδυτές δικαίως θέλουν να ξέρουν πόσο υγιές είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο βάζουν τα λεφτά τους. Οι τράπεζες δεν θέλουν δημοσιότητα για να μην τρομάξουν οι αγορές. Οι, τράπεζες έχουν, οι αγορές με συγχωρείτε έχουν τρομάξει ήδη. Και θα τρομάξουν λιγότερο μόνο με την δημοσιότητα. Και θα ήθελα να ακούσω στην πλευρά των επενδυτών. Αντί να μας λέτε θέλουμε να μείνουν τα πράγματα σταθερά με το να μην ξέρει κανείς τι γίνεται στις τράπεζες. Ας ξεκινήσουμε με εσάς. Να μπω σε ένα-δύο θέματα καταρχάς. Για το δημοσιονομικό θέμα, το μέγεθος του προϋπολογισμού μας, η ΕΣΜΑ, του χρόνου θα έχει, έχει αυξήσει τις προβλέψεις της και ο προπολογισμό που υποβάλαμε στι δημοσιονομικέ αρχές ήταν διαφορετικός από αυτό που είχαμε σκεφτεί αρχικά. Ε, δώσαμε άλλα νούμερα δηλαδή ε, σε σχέση με το 2011. Ο λόγος είναι ότι έκτοτε έγιναν αλλαγές στην νομοθεσία, ε, υπάρχουν νέα νομοθετήματα ε, που μας δίνουν νέε αρμοδιότητες και εξουσίες. Και ακριβώ γι' αυτό ε, προτείνουμε ένα υψηλότερο προπολογισμό για του χρόνου στι δημοσιονομικέ αρχές. Έχει να κάνει με τα καθήκοντα, με τους ελέγχους μας, με το CRA3, με τα επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου, γι' αυτό ακριβώς ε, έχουμε υψηλότερο προπολογισμό. Τι θα γίνει εάν δεν μας δοθούν αυτά τα ποσά. Καταλαβαίνουμε ότι τα πρώτα χρόνια θα περιμένατε ένα έτσι, επιχειρηματικό πνεύμα από εμά και από την ΕΣΜΑ. Δηλαδή να δουλεύουμε σαν τρελή ε, μέχρι να χτίσουμε τον ε, οργανισμό μας. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι τα βασικά που πρέπει να κάνουμε, τα κάνουμε. Το θέμα είναι να προχωρήσει και η Τραπεζική Ένωση. Ε, και οι συζητήσεις που κάναμε την ΕΤΑ, με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, επηρέασαν το, το έργο μας. Εάν δεν μας δοθούν αυτά τα λεφτά, δεν μπορούμε να δουλέψουμε στους διάφορους τομείς και τελικά θα έχουμε, δεν θα έχουμε καλή φήμη. Δεν θα είναι αξιόπιστε οι υποπτικέ αρχέ. Αυτό είναι το πρόβλημα με τι υποπτικέ αρχέ. Είναι σημαντικό δηλαδή να έχουμε καλή φήμη, ε, η δουλειά μα να είναι υψηλή ε, ποιότητα, αν έχουμε ε, αποτυχίες, Αν ξεχάσουμε κάτι, αν κάτι ξεφύγει από εμά, υποδυναμώνουμε, αποδυναμώνουμε το σύστημα. Εάν δεν μας δοθούν αυτά τα λεφτά θα πιεστεί πολύ η οργάνωσή μας. Ε, χρειαζόμαστε 160 λοιπόν. Πάμε τώρα στους καταναλωτές. Στα διαφθομένα προϊόντα κτλ. Τι μπορούμε να πούμε γενικά. Ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι χρηματοπιστωτικοί σύμβουλοι και οι διαχειριστές έχουν αρχίσει να κάνουν αλλαγές. Εστιάζουν περισσότερο στους καταναλωτές αλλά μόλις ξεκίνησαν. Και πρέπει να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ε, στους συμβούλους, στο πώς αντιμετωπίζουν τους ε, πελάτες τους. Να μην τους θεωρούν, ας πούμε, ως ε, ευκαιρίες πλουτισμού. Πρέπει να σκεφτούν πώς μπορούν να τους δώσω τη σωστή συμβουλή και τα, να τους προσφέρω τα σωστά προϊόντα. Πρακτικά πώς γίνεται αυτό. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να εποπτεύουν σωστά τις απαιτήσει που προβλέπει η νομοθεσία, τα MIFID και η ΕΑΚΑ, η ΕΣΜΑ δηλαδή, έχει τον κάνα διολογίας επί της MIFID ε, που θα αναθεωρηθεί από έκθεση ομοτήμων Επίσης, ε, τα ΟΣΕΚΑ είναι προβληματικός τομέας. Και θα ήθελα να ξαναπώ αυτό που είπα προηγουμένως για τα κίνητρα. Έχουμε τώρα μηχανισμό όπου σε πολλά ε, κομμάτια του προϊόντος που πωλείται στον ε, ιδιώτη επενδυτή υπάρχει ένα καθεστώς πληροφόρησης. Ε, θα πρέπει ε, να υπάρχουν προϋποθέσεις καταλληλότητας. Θα πρέπει ε, ο διαχειριστής να συλλέξει ε, πληροφορίες ε, για τον πελάτη. Αν δηλαδή το προϊόν είναι κατάλληλο γι' αυτό. Επανέρχομαι στα κίνητρα. Έχουμε αντικίνητρο, ουσιαστικά, κακά κίνητρα, όπου οι σύμβουλοι δίνουν κίνητρα όταν πουλάνε κάποια προϊόντα και είναι τελείως διαφορετικά από προϊόν σε προϊόν. Ε, δηλαδή τελικά το τα κίνητρα στρεβλώνονται καθοδόν. Αν τα αρχικά κίνητρα δεν είναι σωστά, εμείς δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε. Ό,τι και να κάνουμε ως εποπτικές αρχές. Ε, κάτι που είπα για τις απολαβές των, των υπαλλήλων. Είναι σημαντικό αυτό. Ε, έχει να κάνει με τα κίνητρα. Τα λεφτά στις χρηματαγορές. Όταν δίνει τα λεφτά σου στην τράπεζα τώρα, αντί να έχει κέρδος, πρέπει να πληρώνεις κιόλα. Ποια είναι, ποια είναι η οικονομική λογική, ας πούμε, για αυτές τις δραστηριότητες. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Τώρα, για το θέμα του προϋπολογισμού, να σας δώσω τρία παραδείγματα. Για το τι ισχύει για μας. Καταρχήν ανάλυση των δεδομένων. Κάνουμε πολλέ αναλύσει δεδομένων για τα stress test, για την έκθεση περί που θα πρέπει να σας δώσουμε του χρόνου. Αν δεν έχουμε τους πόρους, θα πρέπει να κάνουμε εξωτερική ανάθεση αυτού του έργου. Τώρα είναι τμήμα των δεδομένων και μην με παρεξηγείτε. Ε, τα διαχειριζόμαστε χάρη στην Bundesbank. Ε, τα διαχειρίζεται για μας γιατί εμείς δεν έχουμε υποδομή πληροφορικής για να το κάνουμε. Το stress test έγινε με πρόγραμμα Excel, δηλαδή ο επιχειρησιακός κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος, βέβαια τελικά όλα πήγαν καλά, ήταν σημαντική πρόκληση, αλλά δείχνει πότε πώς δουλεύουμε και, και η στατιστική μας ικανότητα είναι σχετικά χαμηλή. Οπότε αν θέλουμε σωστή διεκπαιρέωση αυτών των εργασιών χρειαζόμαστε υποδομές ε, και πόρους. Όπως είπα και προηγουμένως υπάρχει θέμα ε, ε, συνάφειας ό,τι αφορά την ε, αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού. Έγιναν κάποιες μαζικές αξιολογίες από ορισμένε χώρες που εμπίπτουν στο, στο μηχανισμό κυρίως αλλά χρειαζόμαστε μία συνάφεια και μία συνοχή. Όσο περισσότερου πόρου έχουμε, τόσο περισσότερη συνοχή μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Όσο λιγότερου πόρου έχουμε, τόσο επαφιόμαστε στι αξιολογήσει των εθνικών αρχών. Τα πράγματα είναι καθαρά και ξάστερα. Τρίτο θέμα, στη θέσπιση των προτύπων, των προδιαγραφών. Το ίδιο ισχύει και εκεί. Όσο λιγότερου πόρου έχουμε, τόσο επαφιόμαστε σε κατάρτιση προτύπων ε, με το μοντέλο των επιτροπών, για παράδειγμα. Οπότε υπάρχουν λιγαρότερε πιθανότητε για γνήσια κοινοτική προσέγγιση και πολύ μεγαλύτερα περιθώρια για εθνική διακριτική ευχέρεια. Σε ό,τι αφορά τώρα την στήριξη των ε, επαυτικών αρχών σε χώρες που υφίστανται πιέσεις ή έχουν υπαχθεί στο, πρόγραμμα της διάσωσης. συμμετέχουμε τώρα σε, προγράμμα, σε αξιολογήσεις της ανακεφαλαίωσης της Ισπανίας και της Κύπρου. Ε, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά ήταν λίγο απογοητευτικό ότι δεν εμπλακήκαμε σε παρόμοια εγχειρήματα και για, σε άλλες χώρες και στην περίπτωση άλλων χωρών. Προσπαθούμε πάντως να συμμετέχουμε με την τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη μας, ιδιαίτερα στα stress test, Αναφερθήκατε στις προνομιούχες αυτές μετοχές της Ισπανίας και τα θέματα του καταναλωτή. Εμείς ε, ε, προσπαθήσαμε να ασκήσουμε επίσης στην Ισπανία για να αναθεωρήσει ε, την νομοθεσία της σε ό,τι αφορά την κατανομή τέτοιων προϊόντων σε μεμονωμένους επενδυτές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τις υποθήκες, το είπα και προηγουμένως, το γεγονός ότι θα εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για τις υποθήκες, για, ε, για τον υπεύθυνο δανεισμό και τη διαχείριση των υπερημεριών είναι σημαντικά θέματα. Βέβαια δεν έχουμε ε, και πολλές ε, αρμοδιότητες από την οδηγία για τα πρότυπα και τους δεσμευτικούς κανόνες. Εμείς μόνο κατευθυντήριες γραμμές μπορούμε να εκδώσουμε ε, πάντως πείτε μας αν σε κάποιους τομείς πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Τώρα σε ό,τι αφορά το φρένο που θα μπει στην Τραπεζική Ένωση. Κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα. Από πέρυσι τον Αύγουστο το προτείναμε ε, ο μηχανισμός χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ο μηχανισμός, ε, ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας να εμπλέκονται άμεσα στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σε άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι σημαντικό να ε, διακοπεί αυτή η σύνδεση με τα κρατικά ομόλογα. Βέβαια αυτή είναι μια βραχυπρόθεσμη λύση και Πιστεύουμε ότι με τη μαζική ανακεφαλοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στον τραπεζικό κλάδο και 13% του ΑΕΠ του κοινοτικού έχει αφιερωθεί στην ενίσχυση του τραπεζικού κλάδου, ελπίζουμε ότι αυτό θα αρκέσει. Στο μέλλον πάντως χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα είναι πολύ πιο θεσμικό κατά τη γνώμη μου και πολύ πιο εύρωστο θεσμικά. Χρειαζόμαστε ελέγχους σε κοινοτικό επίπεδο αλλά και ευθύνε σε κοινοτικό επίπεδο. Δηλαδή να συμβάλλουν και οι τράπεζες σε ένα ευρωπαϊκό ταμείο με ειδικέ εισφορές, ειδικά τέλη και επίσης ε, ε, να είναι αρκετό αυτό και όταν μια τράπεζα ε, χρεοκοπεί να μην αντιμετωπίζει δυσκολίες, να μην αντανακλώνται αυτές οι δυσκολίες στα κρατικά κονδύλια. Πάντως ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν όλοι αυτοί οι πόροι που θα συγκεντρωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά την μακροπροληπτική εποπτεία, εδώ οι, γνώμη, οι απόψεις μου είναι ξεκάθαρες. Μακροπροληπτική εποπτεία σημαίνει έλλειψη ενιαίων κανόνων. Λάθος. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και ενιαίους κανόνες και ελαστικότητα στην εφαρμογή τους ε, και να ε, εφαρμόζονται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε εθνικό επίπεδο ήδη υπάρχουν νέοι κανόνες και τι κεφαλαϊκές απαιτήσει των διαφόρων τραπεζών μπορούμε να τις προσαρμόσουμε στου κινδύνου που έχουν. Αυτό γίνεται με βάση το δεύτερο πυλώνα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο μακροπροληπτικό. Δηλαδή να έχουμε του ίδιου κανόνε και το ίδιο πλαίσιο για το πώ κάθε, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αυξήσει ή να χαλαρώσει κεφαλαϊκά μπάφερ σε ό,τι φορά φούσκες ε, ακινήτων ή φούσκες πιστοτικές και αυτό θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και με σωστό έλεγχο για να μην ε, περιοριστεί η ε, αυτό σε εθνικό επίπεδο, αλλά να, αντιμετωπιστεί το, να αντιμετωπιστούν οι φούσκες. Και αυτό μπορεί να γίνει ε, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις εποπτικές αρχές, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εξασφαλίσει μια γενική επισκόπηση ε, τρόπου εφαρμογή όλων αυτών των εργαλείων. Πάντω, οι κανόνε θα πρέπει να είναι οι ίδιοι και οι μηχανισμοί εφαρμογής τους να προσαρμόζονται στην ε, κατάσταση της κάθε χώρας. Ευχαριστώ για το πρώτο ζήτημα για τον προϋπολογισμό. Και βεβαίως είμαστε σε μια διαδικασία εκτέλεσης και έγκριση σε επίπεδο οδοσού και μετά εμφανίστηκε η Κομισιόν και μας μείωσε τα νούμερα. Πρέπει να είναι σαφές. Αυτό το οποίο εγκρίναμε στο Δουσού ήταν το ελάχιστο δυνατό. Ε, ήδη φτάνοντας στα όρια μας και πάλι σας ευχαριστώ για την στήριξή σας. Ποιες θα είναι οι συνέπειες. Ε, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορούμε να επεκτείνουμε τις ε, δυνατότητες μας και τους πόρους μας και δεν μπορούμε μετά να έχουμε αποτελέσματα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο παραδείγματο χάρη τώρα οικοδομούμε την υποδομή μας ε, την ε, ψηφιακή. Ε, το ανέφερα και στην αλφή. Αν δεν έχουμε αυτούς τους πόρους θα ε, σταματήσει αυτό και θα είναι ε, δυσάρεστο στην πλευρά των ανθρωπίνων πόρων. Χρειαζόμαστε πόρους για αυτή την ανεξάρτητη ανάλυση και πάνω από αυτά βεβαίως τα, τα φυσιολογικά του κανονισμού. Παραδείγματος χάρη τώρα μας ζητάνε και τις αξιολογήσεις ε, της φερεγγιότητας δύο και χρειάζονται γι' αυτό άνθρωποι έμπειροι για να υπάρχει ποιότητα και ανεξάρτητη ανάλυση. Πάντα λέω πως ε, το βασικό περιουσιακό στοιχείο της δικής μου, της αρχής, είναι οι άνθρωποι στους οποίους έχουμε. Και θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια φιλόδοξη διαδικασία όσον αφορά τους καταναλωτές, το ανέφερε ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο για το ζήτημα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και στο επίπεδο της κοινή Επιτροπής και θα ήθελα επί ευκαιρία να αναφέρω και κάτι άλλο. Εγώ υποστηρίζω την σχετική εκπαίδευση. Είναι ξεκάθαρο. Αλλά μην ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι πανάκια. Δεν θα πρέπει το βάρος να μετατίθεται στους καταναλωτές, το βάρος λήψης αποφάσεων δεν πρέπει να θεωρούμε πως θα ε, λάβουν ε, τη λογική απόφαση. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο και το παράδειγμα. Ναι, να δίνουμε καλές πληροφορίες, αλλά πιο συγκρίσιμες, πιο τυποποιημένες. Αυτό προτείνουμε παραδείγματο χάρη στην πλευρά των ατομικών συντάξεων, στην πλευρά της προστασίας των καταναλωτών. Καλύτερες πληροφορίες, όχι περισσότερες, καλύτερες και πιο συγκρίσιμες. Και επίσης ε, και τα κίντρα αυτά τα οποία υπάρχουν, ε, αυτά, οι προμήθειες δηλαδή, είναι σημαντικό κομμάτι και του προϊόντος το οποίο ε, πωλείται και στην οδηγία TRIPS και σε άλλη οδηγία. Εάν μπει αυτό, μπορούμε να βελτιώσουμε κατά πολύ την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει εδώ πέρα ο τρόπος σκέψης υπόδειγμα. Η δημοσιότητα είναι σημαντική, αλλά δεν είναι τα πάντα δεν αρκεί από μόνο της. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια, διεξαγωγή του πώς ε, λειτουργούν οι επιχειρήσεις κτλ. Γιατί μόνο με διαφάνεια δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Ναι, δεν σας βλέπω τώρα. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες αυτές ε, παρουσιάσεις. Νομίζω πως ε, είχαμε μια πάρα πολύ καλή και ποιοτική συζήτηση. Ευχαριστώ και τους Ιερμηνείς. Νομίζω τελειώσαμε στην ώρα μας και μια φορά.